Colleagues, good afternoon. I... Νομίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Την εγκρίναμε, άψογα σας ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω ως πρόεδρος. όσον αφορά την συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου. Να σας πω ότι αυτή η συνεδρίαση διαγράφεται γιατί δεν έχουμε ε, λόγο να συνεδριάσουμε εκτός και αν αλλάξουν τα πράγματα για την ώρα το ακυρώνουμε. Οι συντονιστές όμως αποφάσισαν να διατηρήσουν την συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου στο Στρασβούργο. όπου θα συμπεριληφθεί ψηφοφορία τα benchmarks, καθώς επίσης και για την ετήσια έκθεση. Την 12η Μαρτίου θα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση Econ και Budget. Όπως ξέρετε συζητούμε μαζί υπό, τον, ε, ε, υπό το 25 ε, την, τα μέτρα του κυρίου Γιούνκερ. Όσον αφορά τώρα τις ακροάσεις, έχουμε budget και έκον οι οποίες ε, θα οργανώσουν κοινό, κοινή ακρόαση σχετικά με το πώς μπορεί να καλυφθεί το επιχειρηματικό και επενδυτικό ε, κενό της ε, Ευρώπης. Ε, αυτή η ακρόαση θα λάβει η χώρα στις Βρυξέλλες και θα είναι μια καλή ευκαιρία να συζητηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά ε, το ΕΦΣΥ και θα έχουμε και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, σε μια κοινή συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 5.30 άλλωστε. today we θα έχουμε επομένως ξανά την ευκαιρία να σας δώσουμε όλο το πρόγραμμα εργασίας όσον αφορά το Ταμείο Επενδύσεων. Όσον αφορά τώρα ε, το πιλωτικό πρόγραμμα για, τις, ε, ε, για την για τις ψηφιακές υπογραφές. Νομίζω ότι όλοι τα ξέρετε αυτά, ε, πώς μπορεί να γίνουν αυτές οι υπογραφές ε, με, τη, με τα smartphones και με τις ε, ταμπλέτες. Έχουμε εδώ πολλές ψηφοφορίες. Θα δούμε τώρα μόνο τις τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί από περισσότερο από ένα μέλη. Θα δούμε πώς θα οργανώσουμε τις εργασίες μας. Επίσης, ξέρουμε γενικώ την πιλωτική φάση η οποία την ώρα βασίζεται ε, σε έγγραφα FEC και PDF. Από ό,τι καταλαβαίνω τα προβλήματα τα οποία στην αρχή είχαμε αντιμετωπίσει τώρα δεν υπάρχουν πλέον. Επίσης έχουν υπάρξει ε, προγράμματα κατάρτισης εκπαίδευσης ε, για τους, ε, για τους υπαλλήλους και για τα μέλη. Το ESP δεν είναι υποχρεωτικό αλλά θέλουμε να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει όσοι βουλευτές επιθυμούν να εξακολουθούν να υπογράφουν με τον παραδοσιακό τρόπο μπορούν να το κάνουν και η γραμματεία θα σας ε, ε, δώσει όλες αυτές τις ανακοινώσεις ε, αργότερα μέσα στη βδομάδα. Τέλος, όσον αφορά την, τον τριμερή διάλογο για τις πληρωμές υπηρεσιών, έχει γίνει ο πρώτος τριμερής διάλογος, ο καθένας από, τις, από τους τρεις θεσμούς έχει δώσει τη θέση του έχει, ε, έχει, έχουν συζητηθεί ζητήματα όπως είναι η εποπτεία, όπως είναι η τραπεζική διαμεσολάβηση ε, και τα λοιπά. Έχει δοθεί ούτως ή άλλως ήδη εντολή για να ε, μπορέσουμε να συζητήσουμε επιπλέον και για να δούμε αν και κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα εξέβρεσης πολιτικού συμβιβασμού. Ε, της 2 ε, Μαρτίου 2015 θα λάβει χώρα ο επόμενος τριμερής διάλογος. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω και επομένως μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, σημείο 3 της ημερησίας διατάξεως. Ε, είναι η έκθεση της κυρίας Εύας Καϊλή και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην Εύα, παρακαλώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια από τι βασικέ προτεραιότητε ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο τη ετήσια έκθεση για τη φορολογία φέτο ήταν να μην ακολουθήσουμε ε, μια παράδοση αντιγραφή επικόλυσης. Βλέπουμε στην ετήσια έκθεση φορολογία ότι το Κοινοβούλιο ζητά από το Συμβούλιο επανειλημμένο και από την Επιτροπή τα ίδια πράγματα, αλλά δεν έχουμε δει ικανοποιητικέ βελτιώσει μέχρι τώρα. Εξού και αποφασίσαμε αυτή τη φορά να συντάξουμε μια πιο πολιτική έκθεση. Είχαμε και το σκάνδαλο Lux Leaks, Swiss Leaks και όλα αυτά ζητούν πλέον πολιτική απάντηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να αναλυθεί πολιτική δράση, να τοποθετηθούμε ως πολιτικό όργανο και να μην προσποιούμαστε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα τέτοια έκθεση για τη φορολογία. Είναι το πολιτικό έγγραφο που εκφράσει απόψη Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων Υπήρχαν πάρα πολλές τροπολογίες ε, για το θέμα αυτό, ε, λίξ. καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό και ζητούν την ανάπτυξη πολιτικής δράσης. 300 τροπολογίες συνολικά έχουν κατατεθεί, πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων σε ό,τι αφορά την απονομή κοινωνική δικαιοσύνη, να υπάρχει αυτή η διάσταση στι φορολογικέ πολιτικέ, επίση φορολόγηση κεφαλαίου, πηγών εισοδήματο, ε, μερίσματα, ε, τίτλοι, ε, επιστροφέ αποδόσει ομολόγων και άλλων τίτλων, καταπολέμηση φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή. Επίση, ο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών παραμένει ακροδημοφιλή. Ο πως βλέπουμε τις πολλές τροπολογίες που ζητούν τη βελτίωση και την επέκτασή του. Και τα έσοδα από αυτόν ζητείται είτε να χρησιμοποιούνται για τον, να χρηματοδοτήσουν τον κοινωνικό, κοινωτικό πιοπλισμό ή τις περιβαλλοντικές πολιτικές ή στρατηγικές επενδύσεις. Επίσης, από τις επενδύσεις βλέπουμε ότι οι συνάδελφοί μας ενδιαφέρονται για την εταιρική φορολογία, το CCTB συγκεκριμένα, την φορολογική, την φορολογική βάση εταιριών. Η φορολογία συνδέεται και με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό το βλέπουμε σε διάφορε τροπολογίε. Ή ε, τη μεταχείριση των ΜΜΕ. Υπάρχουν και άλλε τροπολογίε για το φορολογικό ανταγωνισμό. Τέλο. Ξεκολουθεί να υπάρχει μια διχοτόμηση μεταξύ των μελών βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συντονισμό, Αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο LuxLeaks και γι' αυτό πολλοί ζητούν περισσότερη εναρμόση φορολογικών ζητημάτων με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προς, αυτό το σκοπό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ε, είχε δηλώσει και στις προσπάθειες εξέβεσης συμβιβασμού, στηρίζει μια δέσμη πολιτικών για να βοηθήσουμε την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού φόρου φοροδιαφυγής φοροαποφυγή και στηρίζουμε και πολιτικέ για μείωση φορολογικού χάσματος. Επίσης υπάρχει βέβαια κατανόηση τη ανάγκη, ε, να υπάρχει καλή διακυβέρνηση στα φορολογικά ζητήματα, να είναι απλούστερα τα φορολογικά συστήματα και οι φορολογικέ πολιτικές να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και να στηρίζουν τις μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, ε, ως Κοινοβούλιο αναφέρουμε ότι κατανοούμε τις κοινωνικές επιπτώσεις των φορολογικών πολιτικών ιδίων για τους ε, πιο αδύναμους ε, από οικονομικής πλευράς μεταξύ του πληθυσμού. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και κάποια άλλα ζητήματα στο μέλλον για να έχουμε ένα κοινό έδαφος και να χαράξουμε περισσότερες κοινέ πρωτοβουλίες με την ενισχυμένη πλειοψηφία. Βέβαια προ το παρόν υπάρχει επιφυλακτικότητα από κάποια πολιτικά κόμματα. Άρα αυτά τα θέματα που ήθελα να πω ποια είναι. Περιλαμβάνουν τον ορισμό των φορολογικών παραδείσων, τις κυρώσει για του φοροφυγάδε, τι εκθέσει αναχώρα, τη διάβρωση φορολογική βάση, μεταφορά κερδών, BEPS, το FTT, δηλαδή χρηματοπιστωτικό και τη μετατόπιση του φορολογικού βάρου από την εργασία. Ένα επίμαχο θέμα ήταν αυτό με την ταλλαγή πληροφοριών. Για να καταστεί προφανής αυτή η πρακτική τροφολογικών συμφωνιών τύπου tax ruling. Με βάση τις τρέχουσε εξελίξει και την ανησυχία της κοινή γνώμη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει αποφασιστικότητα σε βάρος οποιασδήποτε αδιαφανούς πρακτικής που περιορίζει την ασφάλεια δικαίου διαφορά φορολογουμένου και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Δυστυχώ, βέβαια, υπάρχουν και κάποια ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει κοινό έδαφο, όπω παραδείγματο χάρη για του περιβαλλοντικού φόρου και τέλη, παρότι φαίνεται ότι θα μπορούσαν αυτοί οι φόροι να δημιουργήσουν έσοδα και θέσει απασχόληση και ανάπτυξη, αλλά υπάρχει δυστυχώ πολιτική επιφυλακτικότητα και δισταγμό. τέλο. Υπάρχει το ζήτημα των ε, πληροφοριοδοτών whistleblowers. Όσοι αποκαλύπτουν περιπτώσεις φορολογικής απάτης πρέπει να προστατεύονται και όχι να τιμωρούνται. Παρ' όλα αυτά και τις διαφωνίες δηλαδή που υπάρχουν μπορούμε να πούμε ότι η έκθεση για τη φορολογία φέτος ε, χαρακτηρίζεται από συνεκτικότητα, απλότητα και νομίζω ότι αποτελεί τη βάση για υγιή ε, κοινωνικά υπεύθυνο κοινωνικά υπεύθυνη και σωστή φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ευχαριστούμε την Εύα Καϊλή και τώρα να δώσω το λόγο στο σκιώδη του ΕΛΚ στον κύριο Στόλογιαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την κυρία Καϊλή για τη δουλειά της και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Όχι μόνο με τον σκιώδη του ΕΛΚ, αλλά με όλους τους σκιώδης εισηγητές. Βάσει αυτής της συνεργασίας, με τα χαράς να πω ότι έχουμε δεχτεί τις περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες. Βέβαια, έχουμε πολλές να εξετάσουμε, πολλές συμβαστικές λύσεις. Κάποιες μάλλον, όπου έχουμε κάποια απόκληση στις απόψεις μας. Και θα ήθελα να επισημάνω για την ΆΗ μία έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την εναλλακτική του, ε, φορολογική της φορολογικής βάσης. Δεν ε, υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα της ελάχιστης ενωπημένης βάσης για τις ε, εταιρείε για το ΕΛΑ στο εδάφιο 12B Νομίζω ότι είναι υπέρμετρο να ζητάμε από όλα τα κρατημέλη να προβλέψουν αυτού του είδους την ανάλυση spillover των εθνικών φορολογικών τους πολιτικών, ώστε να αποτιμήσουν τον αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Z είναι μια συμβαστική λύση που τη συζητήσαμε Θέλουμε να καλωσορίσουμε την μετάδοση πληροφοριών όπως αυτές που αποκαλύφθηκαν μέσω του LuxLeaks. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να δώσουμε ένα τέτοιο καλωσόρισμα σε τέτοιου είδους κινήσεις. Δεν είναι καλό να δίνουμε κίνητρα στον κόσμο να κλέβει CD στοιχεία και πληροφορίες με τέτοιους σκοπούς. Επίσης 4 στο ΑΑ. Ο ορισμός της φοροδιαφυγής, της φοροαπάτης, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Νομίζω καλό είναι ο ορισμός αυτός να ε, γίνει από τους επιστήμονες, από τους ακαδημαϊκούς ή έστω από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών. Όταν διάβασα τον ορισμό, πρέπει να σας πω ότι ο ορισμός 4 για τη φοροδιαφυγή και την φοροαπάτη δεν καταλαβαίνω τι διαφορά μπορεί να έχει και να επιβάλλει μεταξύ του νόμιμου και του παρανόμου. Επίσης, θέλουμε χωριστή ψηφοφορία για τις 145, 149 και 247. Όσο για την 145, το δεύτερο τμήμα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, διότι καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει κοινού δεσμευτικού κανόνα για την φορολογία των εταιριών, για να καταπολεμηθεί ο επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και το καθεξής. Εκεί ε, ούτω ή άλλω θα έχουμε μια ειδική επιτροπή πλέον που θα κάνει τι δικέ τη προτάσει για τα θέματα αυτά. Ξεχωριστή ψηφοφορία για την 149, όπω είπα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οποίων και οι αναπτυσσόμενες χώρες για να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Συμφωνούμε με το πρώτο τμήμα της τροπολογίας, αλλά όχι με το δεύτερο. Και για την 247 και πάλι θέλουμε μια ξεχωριστή τροπολογία. Έχουμε ένα πρόβλημα στο πρώτο τμήμα που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει τον σχεδιασμό φορολογική πολιτική στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θεωρούμε ότι όλη η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμεινού είναι ιδιαίτερα ευρεία. Ε, δεν ξέρουμε αν είναι καλή ιδέα να καλέσουμε εμεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει αυτό. Και πάλι ευχαριστώ την κυρία Καϊλή για την πολύ καλή τη δουλειά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα συντηρηθεί και μεταρρυθμιστέ και όντως εισηγητές, ο κύριο Τέρχο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή κυρία εισηγήτρια, Όπω είπα και στι ε, συναντήσει των σκιωδών εισηγητών, Δυστυχώ, η ομάδα του ECR θεωρεί την έκθεση εξαιρετικά δύσκολο να την υποστηρίξει. Καταρχά, το πεδίο εφαρμογή τη έκθεση αυτή πρέπει να είναι πιο επιλεκτικό από ότι Τώρα, η φορολόγηση είναι θέμα των κρατών μελών και εμείς ως ομάδα ECR πιστεύουμε πως έτσι θα έπρεπε να παραμείνει. Και αυτό δεν θα έπρεπε να σας εκπλήσει άλλωστε. Σε γενικές γραμμές πιστεύουμε ότι στο θέμα της φορολόγησης δεν, θεωρούμε, δεν ξέρουμε γιατί θα έπρεπε να δίνουμε συμβουλές στα κράτη-μέλη για φορολογικά ζητήματα. Επίσης, δεν βλέπουμε ε, λόγο ή κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με το τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε πως ο φορολογικός ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι κάτι καλό. Γι' αυτό λοιπόν με δυσκολία θα δεχτούμε τα σχόλια περί συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, συμμεριζόμαστε τα όσα γράφονται για την εθελοντική ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Επίσης, να πω ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε κάποια υποχρεωτική φορολογική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα πλαίσια της κοινή ενωπημένης βάσης φορολογίας εταιριών. Πιστεύουμε πως θα έπρεπε, όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρχει εθελοντική συνεργασία. Επίσης, πιστεύουμε πως η ετήσια έκθεση για τη φορολόγηση είναι πιο πολιτική από ό,τι τις ε, προηγούμενες χρονιές και αυτό είναι κάπως προβληματικό για εμάς, γι' αυτό λοιπόν και με δυσκολία θα το στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου το Κοινοβούλιο απλώς ε, σύμφωνα με τις ε, συνθήκες ε, πρέπει να δώσει την, απο, την γνωμοδότησή του. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, άρα οφείλουμε να δώσουμε και εμείς την πρότασή μας. Θα δώσω τώρα στο Άλντε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλο και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Καηλή γιατί μας έδωσε ε, μια καλή βάση για την ε, έκθεση και την ευχαριστώ γιατί έλαβε υπόψη και τις τροπολογίες μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους άλλους σκιώδεις ε, για την συμβολή τους. Πολλά έχουν υποθεί ήδη τα οποία με αντιπροσωπεύουν. Τώρα, από την προηγούμενη συνεδρίασή μας ε, είδαμε ότι εντωμεταξύ το Κοινοβούλιο αποφάσισε ε, να δημιουργήσει μια εξεταστική επιτροπή η οποία θα μελετήσει ε, τις φορολογικές διευθετήσεις και μέτρα συγκεκριμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να υπάρξουν και συστάσεις για το μέλλον πολύ θετικά βλέπουμε αυτή είναι την Εξεταστική Επιτροπή γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει λόγος ε, και για την επιθετική φορολογική πολιτική αλλά και για τις ε, δυνατότητες και σχέδια φοροαποφυγής ε, που θα αφορούν πολλές χώρες και όχι μόνο μία. Όσον αφορά αυτή την Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε πρόωρα αποτελέσματα. Θα πρέπει να περιμένουμε ε, την εξέταση, τη διερεύνηση η οποία θα λάβει χώρα ε, και μετά αφού θα έχουμε συζητήσει να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Από την άλλη πλευρά και κατά αυτή την έννοια δεν συμφωνούμε με κάποιες τροπολογίες οι οποίες είναι υπερβολικά συγκεκριμένες Συμφωνούμε ωστόσο με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες θα βοηθήσουν ε, την ιδέα της ε, ε, συνολικής αντιμετώπισης των θεμάτων της φοροαποφυγής και της επιθετικής φορολογικής σχεδίασης. Έχουμε πρόβλημα ε, με τις ε, τροπολογίες ε, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στην φορολογική αυτονομία των χώρων μελών π.χ. με περιβαλλοντικούς φόβους, φόρους. Θεωρούμε ότι αυτού του είδους η φορολόγηση θα πρέπει να παραμένει στα χέρια και την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επίσης, σε περίπτωση ε, δηλωμένης, βεβαιωμένης ε, φοροδιαφυγής. Έχουμε κάποιο προβληματισμό όσον αφορά τις κυρώσεις που προτείνονται, αλλά γενικά σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, από την Γκούη Μαρίζα σε ευχαριστώ Ρομπέρτο. Κανονικά δεν είμαι εγώ υπεύθυνη, ο Δημήτρης αλλά δεν είναι εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μου ζήτησε να πάρω τον λόγο ε, και θα διαβάσω το, το σημείωμα που μου άφησε. Θέλουμε και εμείς, λέει ο Δημήτρης, να ευχαριστήσουμε την κυρία Καηλή για την εισηγήτρια, ε, για την ε, καλή συνεργασία, καθώς επίσης και τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Το θέμα της φοροαπάτης και της φοροαποφυγής είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Βρισκόμαστε, θεωρώ, σε θετικό δρόμο, αλλά δεν προχωράει η έκθεση όσο θα έπρεπε Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ε, ε, σωστές γενικές τοποθετήσεις και κάποια μέτρα τα οποία πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά ε, δεν προχωρούν αρκετά. Φοβούμαστε ότι για μία ακόμα φορά θα φτάσουμε σε κάποια γενικόλογα συμπεράσματα και δεν θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τελικά στη ρίζα του. Δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τα νομικά εργαλεία και μέσα έτσι ώστε να καταπολεμήσει την φορά αποφυγή. Όμως μπορεί να πιέσει την Κομισιόν έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα ελέγχου όσον αφορά τις εμπορικές διεθνείς δραστηριότητες ε, των εμπορικών εταιριών, τους, τις offshore εταιρείε, ε, καθώς επίσης ε, και τους φορολογικούς παραδείσους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορθά οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, δημιουργώντας μια εξεταστική επιτροπή η οποία πραγματικά θα μπορέσει σε βάθος να μελετήσει το θέμα. Θα πρέπει ε, τα συμπεράσματα, ε, οι εργασίες της Επιτροπής να είναι δημόσιες, να δημοσιοποιηθούν και τα συμπεράσματα να είναι συγκεκριμένα. Τώρα, όσον αφορά τις προτεραιότητες, ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα ε, να ε, μεταφερθεί το φορολογικό βάρος στον πλούτο να, και να δημιουργηθούν με τον τρόπο αυτό σωστής ποιότητας θέσεις εργασίας. δεύτερον, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συνολική στρατηγική έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ε, οι διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες ε, καθώς επίσης και τα κέρδη τα οποία ε, έχουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Τρίτον, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των φορολογικών παραδείσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέταρτον, θα πρέπει να ενισχυθεί η φορολογική συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρώπης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την φοροαπάτη και την φοροαποφυγή αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει αυτά να ενταχθούν σε μία μακροχρόνια ε, πολιτική χρειάζονται φορολογικές πολιτικές ε, βάσει των οποίων θα κατανεμηθεί ο πλούτος και το βάρος σωστά ε, και να μην είναι οι εργαζόμενοι οι μόνοι που πληρώνουν φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Μαρίζα από τους πράσινους η μόνη καμκάτω. I'd like to echo Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καλή και όλους τους σκιώδες εισηγητές. Είχατε δίκιο κυρία Καλή, ήταν μια πάρα πολύ περίπλοκη έκθεση με πολλές τροπολογίες. Η δική μου τοποθέτηση είναι καταρχάς να καλωσορίσω τα όσα είπαν οι ε, προηγούμενοι εισηγητέ για την αντιμετώπιση τη ε, φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη, αλλά και για την ανάγκη επενδύσεων για την κοινωνία. Φυσικά ω πράσινη Είμαστε απογοητευμένοι για την ε, έλλειψη μέτρων για την βελτίωση της πρόσβασης στα έγγραφα. Ωστόσο, καλωσορίζουμε το γεγονός της δημιουργίας αυτής της ειδική Επιτροπής αυτήν την εβδομάδα και θα ε, συνεργαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για το έργο τους. Επίσης, πιστεύω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε ε, τα πράγματα. Η φορολόγηση μας επιτρέπει να χρηματοδοτήσουμε δημοσιονομικούς ε, στόχους αλλά και να δώσουμε κίνητρα και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείε να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο και συμπεριλαμβάνονται και τα ε, περιβαλλοντικά ζητήματα σε αυτό. Πιστεύω πως η πολιτική μας πρέπει να έχει στόχους την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση που έχουμε στην φοροαποφυγή. Είμαι ωστόσο πεπισμένη ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε πρόοδο στο θέμα αυτό σε αυτή τη θητεία. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον στρατηγικό ρόλο που έχει η φορολόγηση. Η φετινή χρονιά θα τελειώσει με τις ε, πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις στο Παρίσι. Και δεδομένου τούτου δεν πιστεύω πως έχει δοθεί αρκετή έμφαση στην ε, περιβαλλοντική και ενεργειακή φορολόγηση στην έκθεση αυτή. Πιστεύω πως δεν πρέπει να αφήσουμε το λόμπι των ορυκτών καυσίμων να υπερισχύσει και πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου. Thank uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Άνεμανς, έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στην τέση έκθεση για τη φορολογία γίνεται λόγο ε, για παγκόσμια πρότυπα διοικητική συνεργασία. Υποτίθεται ότι καταρτίζονται αυτά τα πρότυπα και όλα ωραία και καλά ακούγονται. Τι θα γίνει όμως μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου πριν από λίγες μόλις ημέρες στα πρωτοσέλιδα ε, αναφέρονταν αυτές οι φορολογικές συμφωνίες τύπου tax ruling με κάποιες πολυεθνικές. Άρα ακόμα πάρα πολύ νοπό το ζήτημα αυτό leaks. τι θα γίνει όταν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Κάποιες φορές ε, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης ε, της ε, φοροδιαφυγής με κάποιες φορολογικές συμφωνίες όταν είναι μεγάλο το βάρος ε, στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Αναζητούνται λοιπόν χώρες με καλύτερες συνθήκες και αναζητείται η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων. Ωραία, μιλάμε για βάρος που βαρύνει αυτές τις επιχειρήσεις. Τι θα γίνει όμως μετά. Θέλουμε να έχουμε παντού τον ίδιο ΦΠΑ. Έχουμε όμω διαφορετικού συντελεστέ ε, φορολογικού από τη μια χώρα στην άλλη και από τον ένα κλάδο στον άλλο. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα τα βάλουμε όλα ε, στο ίδιο επίπεδο, θα τα εξομοιώσουμε όλα. Μήπως θα πρέπει πρώτα απ' όλα η ειδική επιτροπή να εξετάσει τα σχετικά ζητήματα ο Γιουνκέρ και ο Φερχόφστατ ε, θέλουν ε, την Ομοσπονδία Ευρώπη. Δεν την ελάμβαναν όμως τόσο σοβαρά όταν τα πρωθυπουργοί. Thank you. Η συγγήτρια παρακαλώ για κάποιες τελικές παρατηρήσεις. As you see, uh, Βλέπετε ότι συμφωνούμε με τα περισσότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Σας είπα ότι είχαν υποβληθεί 300 τροπολογίες, προσπαθήσαμε να έχουμε κάποιους συμβιβασμούς, υπάρχουν όμως θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν άμεσα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνεισέφεραν παραγωγικά με τις τροπολογίες τους στην έκθεση και όχι μόνο με τις τροπολογίες τους αλλά και με τις υποδείξεις και τις προτάξεις τους και θέλω να ευχαριστήσω και τους κοιόδους συζητητές. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία μαζί τους για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης και τους παρακαλώ να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και στο μέλλον. Άλλωστε, περισσότερο θα είμαστε μέλη και της Ειδικής Επιτροπής. Θα μπορέσουμε λοιπόν με περισσότερη λεπτομέρεια και από πιο κοντά να παρακολουθήσουμε τη δουλειά. Αυτό θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον Μάρκο και τον Μπενουά, τους εμπειρογνώμονες μας από την Γραμματεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα, γίνει ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εργασία της, στην εισηγήτρια, αλλά και τους ε, ε Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Έχουμε μια μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη και θα πάμε στον κύριο Σόρου, στην έκθεση του κυρίου Σόρου σχετικά με την διαφάνεια των και την ασφάλεια ε, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Κύριε Σόρου, παρακαλώ. I will keep it in my mind. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ και τους κοιόδης ηγητές. Πριν από μερικές εβδομάδες ως εισηγητής ε, είχα παρουσιάσει τις πρώτες μου ιδέες σχετικά με την διαφάνεια ε, των ε, συναλλαγών ε, και είχα έρθει σε επαφή και με τους ε, ε, σκιώδεις και είχα πάρει και κάποιες ιδέες από την Κομισιόν. Αποφασίσαμε να επιμηκύνουμε την προθεσμία υποβολής τροπολογιών όπως ζητήθηκε. Βεβαίως δεν θα διαφοροποιηθεί η χρονολογία που έχουμε επιλέξει και το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την νομοθετική αντιμετώπιση. 150 μέχρι τώρα είναι οι τροπολογίες τις διάβασα πολύ προσεκτικά. Ακόμα πιο προσεκτικά μάλιστα έχω διαβάσει τις τροπολογίες οι οποίες έχουν από κοινού υποβληθεί από πολλούς ε, σκιώδης και που θεωρώ ότι εκφράζουν ε, μεγάλο τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, οι αναφέρονται ε, και σε θέματα τα οποία δεν είχαμε με όλες τις πολιτικές ομάδες τη δυνατότητα να συζητήσουμε γιατί δεν είχαν όλοι ε, αναθέσει την σκιώδη αντιμετώπιση της ε, έκθεσης. Ε, εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει κάποια απόσταση, ωστόσο είμαι, ε, έχω εμπιστοσύνη, είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να μειώσουμε την απόσταση αυτή. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε πιθανές συμβιβαστικές λύσεις και θα έχουμε μάλιστα στη διάρκεια της εβδομάδας μια συνάντηση με τους σκιώδεις έτσι ώστε να διαλευκάνουμε κάποια σημεία Τώρα, διαβάζοντας ε, τις ε, τροπολογίες, να πω ποια είναι τα σημεία τα οποία φαίνεται να είναι πιο σημαντικά. Το άρθρο 2 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Ήδη συζητήθηκε το θέμα αυτό και νομίζω πάντως ότι χρειάζεται να εμβαθύνουμε περισσότερο. Ε, δηλαδή, το βασικό στοιχείο είναι εάν θα πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις ε, όσον αφορά τις κεντρικές τράπεζες και σε σχέση συγκεκριμένα με την υποχρέωση αναφοράς και διαφάνειας. Στην προηγούμενη συζήτηση αναφέρθηκε ότι οι απαιτήσει του απορρίτου ε, των νομισματικών πολιτικών που ε, διεξάγουν οι, ευρωπαϊκές, ε, οι, οι κεντρικές τράπεζες μπορεί εν μέρη να δικαιολογούν αυτήν την εξαίρεση από την υποχρέωση αναφοράς και διαφάνειας. Μελέτησα το θέμα και θεωρώ ότι η στάση αυτή μπορεί να γίνει δεχτή. Ωστόσο, υπήρξαν και διαφορετικές ε, ε, σκέψεις ε, οι οποίες μας οδηγούν στο να μελετήσουμε περισσότερο το θέμα αυτό όσον αφορά συγκεκριμένα τις ε, συναλλαγές ε, οι οποίες αυτού του είδους οι τράπεζες ε, κάνουν. Είναι πολλές οι πολιτικές ομάδες οι οποίες συζητούν πολύ το θέμα. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μια χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάγκη διαφάνειας από τη μία και στην ανάγκη της συγκεκριμένης απόρριτης πολιτικής που μπορεί να έχουν οι τράπεζες αυτές. Κατά αυτή την έννοια έχει υποβληθεί η τροπολογία 215, έχει κλείσει το μικρόφωνο του ομιλητού, δεν τον ακούμε. Το άρθρο 3 τώρα. Το άρθρο 3 ασχολείται με τους ορισμούς. Και εδώ θα πρέπει ίσως ε, να μελετήσουμε σε βάθος ε, κάποια θέματα, κυρίως όσον αφορά τα νομικά ζητήματα, τα οποία ε, ίσως δημιουργούν πρόβλημα όσον αφορά κυρίως ε, την δυνατότητα να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ή διαιτησία. Η δυνατότητα λοιπόν ε, να ξεφύγει κανείς από τον ε, ε, κανονισμό μέσα από μονοπάτια τα οποία δεν είναι πάντα τα καλύτερα. Πιστεύουμε ότι και εδώ μπορούμε να φτάσουμε σε μία λύση η οποία θα ρυθμίζει αυτήν την διαιτησία με τρόπο αποδεκτό από όλους. Άρθρο 4 που αναφέρεται στην ε, έκθεση και τη διαφάνεια. Υπάρχουν εδώ πολλές τροπολογίες ε, τις οποίες θα μελετήσω. Μερικές όμως από αυτές τις τροπολογίες μου φαίνεται ότι πολύ δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν. Δηλαδή ε, κυρίως εκεί που εκτός από την έκθεση, την υποβολή έκθεσης αναφέρεται και το, η δυνατότητα μεταβίβασης νομικών εξουσιών. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία τα οποία αφορούν τα άρθρα 20 και 21. Επ' αυτών των άρθρων έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες. Οι διαφορές βέβαια είναι ε, μικρές. Όσον αφορά το άρθρο 28 για την θέση σε ισχύ, εδώ προτείνεται μία πιο βαθμιαία προσέγγιση ναι, δηλαδή σιγά σιγά να εφαρμοστεί το νομοθέτημα αυτό και όχι ε, ολόκληρο, όχι το σύνολό του σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχει πάντως ένα σημείο το οποίο είναι πιο περίπλοκο και που αφορά ε, την ε, εξαίρεση για τις περιπτώσεις του Transfer Collective Agreement. Αναφέρομαι κυρίως στην τροπολογία 204. Εδώ δεν είμαι πάρα πολύ ευτυχής με όλα αυτά, γιατί πιστεύω ότι εάν γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία, τότε ε, θα περιορίσουμε πάρα πολύ την αγορά γιατί 95% των συναλλαγών γίνονται βάσει αυτού του Titan Transfer Agreement επομένως εδώ πιστεύω ότι θα έχουμε δυσκολία, γιατί στην ουσία θα διαγραφεί το μεγαλύτερο κομμάτι της, ε, ε, του, του νομοθετήματος αυτού. Ε, εν πάση περιπτώσει θα ξανασυζητήσουμε και θα δούμε. Όσον αφορά τώρα τα haircuts, όσον αφορά τα κουρέματα, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Ξέρετε και θα θυμάστε φαντάζομαι ότι στο αρχικό μου προσχέδιο είχα ε, εισαγάγει αυτές ε, τις τροποποιήσεις ας πούμε στο 15 αναλύοντας και τις τροπολογίες και λαμβάνοντας υπόψη και τις συζητήσεις, βλέπω ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός. Από τη μία πλευρά η Γκουε, η Πράσινη, η δικιά μου ομάδα, ένα κομμάτι του FDD θεωρούν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν κάποιες διατάξεις για τα κουρέματα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τους συναδέλφους Άλντε, ΕΛΚ, που θέλουν παραπομπή αυτής της απόφασης σε άλλη σε άλλο νομοθέτημα πέρα από τις διαφορές οι οποίες είναι σαφείς πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα προσέγγισης από την αρχική θέση. Δεν συζητάμε πλέον για το εάν και κατά πόσον θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο για τα κουρέματα αλλά οι μεγάλες διαφορές αφορούν το χρονοδιάγραμμα ε, βάσει του οποίου κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση, μπορούν να γίνουν περαιτέρω ε, βήματα πρόοδου και ενδεχομένως να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό. Τώρα θα αφήσω να, να μιλήσουν ε, οι σκιώδεις εισηγητές, οι συνάδελφοι, τους οποίους βεβαίως ευχαριστώ για την διαθεσιμότητά τους, για τη συνεργασία τους, για την καλή δουλειά που κάναμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Ρενάτο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Τανούτα Χιούπνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να πω ότι ο κανόνας αυτός δεν είναι ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων. Είναι ένας κανονισμός για την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις ε, συναλλαγές αυτές και για τη διαφάνεια. Μερικά από τα προβλήματα που μπορεί ακόμη να αντιμετωπίζουμε στη διαδικασία εξέτασης και αναζήτησης συμβαστικών λύσεων αυτά μπορεί να οφείλονται, οι δυσκολίες μπορεί να οφείλονται στο ότι Κάποιοι από του συναδέλφου που είναι μέλη τη Επιτροπή αυτή θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία για να καλύψουν περισσότερα ζητήματα πέραν αυτών των δύο που μπορούμε ε, χωρίς πρόβλημα να επιλύσουμε στο πλαίσιο αυτής της πρότασης. Είμαι πιο αισιόδοξη από το Ρενάτο ως προς το δυναμικό για την εξέβρεση συμβαστικών λύσεων. και περιμένω να δω την τελική εκδοχή των συμβιβαστικών προτάσεων που θα προβληθούν. Υπάρχει σαφές, σαφές δυναμικό ε, και σαφής δυνατότητα να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ μας. Να θίξω αρκετά ζητήματα που ήθελα να καλυφθούν από τις τροπολογίες μου ή από τις τροπολογίες που επεξεργαστήκαμε με μερικούς από τους συναδέλφους. Και να ευχαριστήσω καταρχάς τον Ρενάτο που συμφώνησε μαζί μου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το γεγονό ότι θα πρέπει το άχθο για τι μικρομεσαίε να ελαφρυνθεί. Θα πρέπει και αυτέ να καλύψουν τι απαιτήσει υποβολή εκθέσεων για τι ε, συναλλαγέ του χρηματοδότηση τίτλων με του αντισυμβαλωμένου και εκεί θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση. Εξαίρεση για τι μικρομεσαίε υπό την έννοια ότι θα είναι υποχρέωση του αντισυμβαλωμένου να υποβάλλει πληροφορίε για τι συναλλαγέ αυτού του είδου με τι μικρομεσαίε. Τώρα για του ορισμού. Χρειαζόμαστε ορισμού ε, πιο σαφεί και κάποιοι έτσι αλλιώ λείπουν από τον κανονισμό, οπότε προσέθεσα τρία ή τέσσερα σημεία για τους ορισμούς όπου ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Ε, ακόμη για την εξονοχιστική λεπτομέρεια της υποβολής εκθέσεων. Το θέμα των ε, εκθέσεων που θα πηγαίνουν στην ΕΣΜΑ ή στις ε, εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να ε, έχουν επαρκές επίπεδο λεπτομέρεια, όμως οι πληροφορίες πηγαίνουν και στους φορείς της λιανικής αγοράς. Εκεί χρειάζεται άλλο επίπεδο λεπτομέρεια. Ε, αυτή η διαφοροποίηση νομίζω είναι δικαιολογημένη. Για τα κουρέματα ε, θα συμφωνήσουμε. Ίσως να παραμείνει ο διχασμός αυτός μέχρι τέλους, γιατί κάποιοι από εμά θέλουμε να διαθετηθούν τα κουρέματα και κάποιοι άλλοι όχι. Και κάποιοι πιστεύουμε ότι βάσει των πληροφοριών που διαθέτουμε και βάσει του συστήματος δεν μπορούμε με αυτόν τον κανονισμό να λύσουμε το θέμα των ε, κουρεμάτων, των χέκατς. Γι' αυτό ε, ευθύ εξ αρχή ε, με τη ρήτρα αναθεώρηση ήμουν συμφωνή ώστε όπως άλλοι συνάδελφοι προτείνουν μαζί και εγώ μετά από 18 μήνες από τη θέση σχέση του κανονισμού η ΕΣΜΑ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να υποβάλουν έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τελικό συμπέρασμα του πώς επηρεάζονται πώς επηρεάζονται αυτές οι συναλλαγές από τον συγκεκριμένο κανονισμό και με τα παράγωγα προϊόντα και με τι παράπλευρε συνέπειε. Θα πρέπει μετά η Επιτροπή να υποβάλει μια σωστή πρόταση για τα κουρέματα, διότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και ένα, και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να παράσχουμε ασφάλεια και στου συναλλασσομένου στην αγορά. Επίση για την επαναχρησιμοποίηση. Εκεί Νομίζω πρέπει επίση να εξευρεθεί τροπολογική λύση. Τώρα, η δική μου ερμηνεία των όσων προτείνει ο Ρενάτο είναι ότι για τι παράπλευρε συναλλαγέ για τις για τις συναλλαγές εξασφαλίσεων θα πρέπει να προβλεφθεί κάτι σχετικά και για την μεταφορά τίτλων και τις σχετικές εξασφαλίσεις που θα συναρτώνται σε αυτές τις συναλλαγές εκεί κάτι θα πρέπει να προβλεφθεί και να έχουμε μια τέτοια διατύπωση που θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε τον κίνδυνο οι εξασφαλίσεις να μην εξαρτώνται από την ενδεχόμενη πτώχευση του ε, εξασφαλίζοντα. Σήμερα λοιπόν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα διακρίνουμε αυτά και συζητήσαμε και με άλλους σκιώδεις το θέμα της δυνατότητας, οι θέσεις να καλύπτονται και αυτές από την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, όχι μόνο οι συναλλαγές οι ίδιες, δηλαδή για το margin lending και το securities lending θα πρέπει και εκεί να υπάρξει μια καταγραφή των στοιχείων και μια υποβολή έκθεσης. Υπάρχει και το μεγάλο θέμα της ε, μονής ή της διπλής έκθεσης. Εκεί θα πρέπει να ε, δούμε τι θα κάνουμε και τι θα επιλέξουμε, γιατί επιχειρήματα υπάρχουν υπέρ και του ενός και του άλλου. Και για τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους ξέρουμε τι ισχύει και γι' αυτό η συμβιβαστική λύση που θα βρεθεί θα πρέπει να προκύψει για τη δυνατότητα οι αντισυμβαλόμενοι σε μια συναλλαγή να μπορούν νομικώς να εκχωρήσουν την υποχρέωση που έκθεση σε έναν από τους ε, αντισυμβαλωμένους. Ε, με πλήρη σεβασμό λοιπόν του νομικού πλαισίου θα είναι μια δέσμευση νομική αυτή και θα υπάρχει και ε, ασφάλεια και βεβαιότητα. Ε, ανεξαρτήτως όμως πιστεύουμε ότι η ΕΣΜΑ θα σκεφτεί στο μέλλον να επιβάλλει περισσότερες υποχρεώσεις ε, έκθεσης. Διότι σε κάποιες περιπτώσεις η διπλή υποβολή είναι απαραίτητη. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μάλλον στο μέλλον. Και επίσης παραμένει και το θέμα του κατά πόσον ο κανονισμός αυτός θα τεθεί σε ισχύ με μια ε, ε, προσέγγιση σταδιακής εξάλληψης σταδιακή κατάργηση. Αυτή η διαδικασία νομίζω ότι μπορεί να καλύπτεται από κατεξουσιοδότηση πράξη. Αυτά ήταν τα βασικά σχόλια που ήθελα να κάνω οπωσδήποτε, γιατί εκεί πιστεύω ότι υπάρχουν ζητήματα. Ένα ζήτημα που δεν πρόλαβα να αναφέρω είναι οι κεντρικέ τράπεζε και το τι θα κάνουν εκείνες με την υποβολή εκθέσεων. Εκεί υπάρχουν πολλά επιχειρήματα και υπέρ και κατά. Νομίζω ότι μια συμβαστική λύση αρχίζει να διαφαίνεται ε, στις συζητήσεις μας και ελπίζω ότι θα την ε, ολοκληρώσουμε, ώστε να έχουμε μια σαφή νομισματική πολιτική, ασφαλή νομισματική πολιτική και να παρέχονται και απαραίτητε πληροφορίε ταυτόχρονα. Για ένα μεγάλο τμήμα των ε, συναλλαγών χρηματοδότηση τίτλων, όπου ε, εμπλέκονται οι κεντρικέ τράπεζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ, Ντανούτα. Η Κέι Σουίνμπορν δυστυχώ δεν είναι εδώ σήμερα, οπότε θα δώσω το λόγο τώρα στον συναδέλφο από το ECR. Σα ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Κέι Σουίνμπερν, η οποία δυστυχώς είναι άρρωστη και δεν μπόρεσε να έρθει. Θα μιλήσω λοιπόν εκ μέρους της. Η κυρία Σουίνμπερν χαίρεται γιατί υπήρξε συμφωνία μεταξύ σχεδόν εισηγητών για σχεδόν όλα τα ζητήματα του φακέλου αυτού. Οι τροπολογίες μας στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με την βελτίωση της προσέγγισης και με μικρές λεπτομέρειες. Όσον αφορά την αποκάλυψη και την υποβολή εκθέσεων, η κυρία Σουίνμπορν θα ήθελε να δοθεί έμφαση στο διοικητικό φόρτο που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείε με τι ε, νέε απαιτήσει που θα εισαγάγει ο κανονισμό αυτό. Καταρχά, θα πρέπει να καταστεί σαφέ ότι θα είναι δυνατόν να δοθεί σε άλλον αντισυμβαλόμενο υποχρέωση υποβολή εκθέσεων. Όσον αφορά τους μη ε, χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλαιόμενους που δεν έχουν την δυνατότητα υποβολής εκθέσεων. Επίσης, υπάρχουν νέες ε, απαιτήσει για την ε, αποκάλυψη στοιχείων οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και θα μπορούμε να αντλήσουμε από το έσμα γι' αυτό. Η κυρία Σουίνμπερν επίσης δεν θα ήθελε να ποινικοποιηθούν εκείνα τα ταμεία που ήδη έχουν υψηλά ποσοστά ε, αποκαλύψεις πληροφοριών. Επίσης, η κυρία Σουίνπον θα ήθελε να δει μια συνεκτική προσέγγιση που θα συνδυάζει και άλλα νομοθετήματα και θα χρησιμοποιεί το εφιστάμενο πλαίσιο για, ε, της ε, οδηγίας για υποβολή ε, εκθέσεων μη χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα. Τώρα, όσον αφορά τους ε, ορισμούς, η κυρία Σπίνμπορν έχει ήδη αναφέρει σε προηγούμενες συναντήσεις ότι παρότι συμφωνεί με πολλούς από τους ορισμούς, προτείνει ελαφρές βελτιώσεις και τροποποιήσεις έτσι ώστε να διευκρινιστεί καλύτερα ε, να διευκρινιστούν καλύτερα οι ορισμοί. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί σαφήνεια, χωρίς όμως να τεθεί υπονομική αμφισβήτηση ε, οι συναλλαγές εξασφαλίσεων. Επίσης, η κυρία Σφίνπερν επιθυμεί να αποδοθεί περισσότερη νομική ασφάλεια στους ορισμούς. Τώρα όσον αφορά τα κουρέματα στα στα περιθώρια. Χρειάζεται ακόμα να περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος πρώτο τοποθετηθούμε και επίσης πρέπει να υπάρχει σύγκληση με μια εν γέννη βελτιωμένη προσέγγιση. Τέλος, η κυρία Σουίνπορν θα ήθελε να ζητήσει να δοθεί περισσότερη προσοχή τις ημερομηνίες και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής για τα ρυθμιστικά πρότυπα. Ε, κανονισμοί όπως η CSTR και ο MIFID έχουν δεχθεί κριτική από την ΕΣΜΑ γιατί χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γίνουν οι κατάλληλοι τεχνικοί έλεγχοι. Επίσης, το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει ενδελεχώς πάρα πολύ μεγάλο όγκο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και η κυρία Σουίνπορν έχει υποβάλει πρωτοβουλίες, ε, τροπολογίες, με συγχωρείτε, για ένα, ε, για περισσότερο χρόνο εξέτασης των λεπτομεριών, έτσι ώστε και η ΕΣΜΑ να έχει περισσότερο χρόνο να αξιολογήσει την ποιότητα των εργασιών, αλλά και το Κοινοβούλιο να καταφέρει να εξετάσει με προσοχή όλες τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Επίσης, συμφωνούμε όλοι ότι η δουλειά μας εδώ είναι ε, να διασφαλίσουμε ότι με, την δικιά, με το δικό μας αυτό θέτημα θα αποφευθούν οι συστημικοί κίνδυνοι και ε, θα γίνουν διαφανείς κάποιες συναλλαγές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός τραπεζικής εποπτείας. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε και η κυρία Χούμπνερ προηγουμένως, δηλαδή ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια σημαντικά στοιχεία. Ένα, ότι θα πρέπει να αφήσουμε ως έχουν οι αγορές οι οποίες λειτουργούν καλά χωρίς να τις επιβαρύνουμε. Δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς γιατί είναι τεχνικός ο φάκελος. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν σαφείς για τις νομικές επιπτώσεις. Τρίτον, να μην κάνουμε ε, να μην παρεμβούμε, παρέμβουμε κατά κάποιο τρόπο ε, σε ε, εργασίες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Κατά τα άλλα θα συμφωνήσω και με τους συναδέλφους που μίλησαν προηγουμένως. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπαν. Υπάρχουν κάποια στοιχεία όμως τα οποία θα ήθελα εδώ να αναπτύξω δικά μου στοιχεία. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τα κουρέματα, haircuts. Εδώ δεν είναι να πει κανείς ναι ή όχι, συμφωνώ, διαφωνώ. Νομίζω ότι εδώ χρειαζόμαστε καλή διακυβέρνηση έτσι ώστε να υπάρχει σωστή πληροφόρηση όσον αφορά τα κουρέματα. Επίσης το θέμα της χρονικής στιγμής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε άποψη χωρίς να έχει γίνει ε, μελέτη αντικτύπου. Δεύτερον, ε, μιλάμε εδώ για παγκόσμιο συνολικό ε, εμπόριο και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε ε, οι εργασίες να είναι ταυτόχρονες και συμβατές. Τρίτον, μιλάμε για μία βαθμιαία ε, εφαρμογή των απαιτήσεων ε, ε, υποβολής εκθέσεων. Θα πρέπει η ΕΣΜΑ πάντως να αποφασίσει τι είδους ακριβώς θα είναι οι εκθέσεις αυτές και σε ποιο βαθμό λεπτομέρειας θα φτάνουν. Αυτό θα το δούμε στις επόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά τώρα την διαφάνεια Έχουμε υποβάλει μια τροπολογία έτσι ώστε να αποφευχθεί η, ε, το υπερβολικό διοικητικό άχθος για τις ε, επιχειρήσεις. Θα πρέπει βεβαίως να εισάγουμε στοιχεία τα οποία εν τέλει ε, θα είναι εποφέλη Η ΕΣΜΑ θα πρέπει να μελετήσει και τις παρούσες διατάξεις όσον αφορά όλα τα τραπεζικά προϊόντα. Αυτά ήθελα να πω, αλλά και ένα τελευταίο ακόμα, το οποίο θα ήθελα να θίξω. With definitions. Uh, ε, κάποιες ε, αντίθετες ε, από το προσδοκόμενο επιπτώσεις Κατά αυτή την έννοια πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, είμαστε πάρα πολύ ε, προσεκτικοί όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και όσον αφορά τους ορισμούς, ε, οι οποίοι οι ορισμοί δεν θα πρέπει να αφήνουν κανένα περιθώριο νομικής ασάφειας. Θα πρέπει να μελετήσουμε εκ των προτέρων ε, την ε, νομική επίπτωση όλων των προτινομένων μας ε, ας πούμε όσον αφορά αυτό το title and title transfer που αναφέρατε προηγουμένως θα πρέπει να δούμε πριν καταλήξουμε σε κάποια συγκεκριμένη πρόταση να δούμε λέω ποιες θα είναι οι νομικές επιπτώσεις και αυτό να γίνει με όλες τις προτάσεις που κάνουμε νομίζω ότι αυτό που θέλουμε είναι ένα σαφές πλαίσιο για τις Μελλοντικέ τραπεζικές συναλλαγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Φίλιπ Τεμπάκερ. Η κυρία Κάρη έχει το λόγο για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Σόρου. Ακούσαμε μια πολύ καλή εισαγωγή και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε ότι αφενός θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζουμε τους κινδύνους με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, αλλά θέλουμε και κάτι παραπάνω την άλλη πλευρά, δηλαδή να δούμε και να ρυθμίσουμε πώς χρησιμοποιούνται. Δηλαδή θέλουμε διαφάνεια, αλλά και κανόνες για την χρήση των συναλλαγών αυτών. Σας στηρίζουμε λοιπόν στις προτάσεις σας. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες ομάδας μας, ομάδας GoNGL με τις οποίες δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε άρδιν την κατάσταση, αλλά να διευκρινίσουμε λίγο παραπάνω ακριβώς τι γίνεται. Με στόχο μας τη μείωση των συστημικών κινδύνων έξω και προτείνουμε περιορισμό των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης, να γίνεται άπαξη η επαναχρησιμοποίηση. Το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό. Δεν θέλουμε να μην υπάρχει καθόλου αυτή η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, αλλά να μπορεί να γίνει μόνο μία φορά. Όταν μιλάμε για τη ρύθμιση του κουκουρέματος, ε, Χέρκατ, ε, συμφωνώ. Ε, μάλλον χαίρομαι που συμφωνεί και ο εισηγητής, αλλά σίγουρα χρειάζονται κανόνες. Ακόμη και αν δεν έχουμε ακόμη πλήρες συστάσεις από την ΕΚΤ, εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει με υπευθυνότητα ήδη να ξεκινήσουμε να καταρτίζουμε σχετικές ρυθμίσεις. Έχουμε τη βάση, δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και να μην προσπαθήσουμε ήδη από τώρα να ρυθμίσουμε τα κουρέματα. Εναλλακτική βέβαια θα ήταν να περιμένουμε και να ολοκληρώσουμε τους νέους κανόνες μόνο αφού πάρουμε στα χέρια μας τις συστάσεις της ΕΚΤ. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι στηρίζουμε την ένταξη της ΕΚΤ στον κανονισμό αυτό, διότι δεν θέλουμε πολλά παραθυράκια, θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια. Δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε γιατί η Κεντρική Τράπεζα φοβάται τόσο πολύ να δώσει τα στοιχεία αυτά. Δεν λέμε να τα δημοσιοποιήσει για όλους, αλλά για τις κυβερνήσεις, για τα θεσμικά όργανα. Δεν θέλουμε να υπάρχουν λοιπόν παραθυράκια. Κατά τα λοιπά νομίζω ότι έχουμε μια καλή βάση συμβιβασμού και περιμένω τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σκοτ, κάτω για τους πράσινους, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συγγνώμη για από την κυρία Εύα Ζολή που βρίσκεται σε αποστολή και δεν μπορεί να είναι εδώ. Είχε κάποια τεχνικά σχόλια και θα τα κάνω εγώ εκ μέρου τη για αυτό το πολύ τεχνικό θέμα. Καταρχά, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Σόρου, για τον πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή του κάποια σημεία που ε, συνάδουν με τον κανονισμό. Είμαστε υπέρ των ελάχιστων προτύπων για την ε, αξιολόγηση των εξασφαλίσεων και των σχετικών προτύπων και θα πρέπει και τα μη χρηματιστηριακά στοιχεία, τα μη χρηματοπιστωτικά μάλλον στοιχεία να καλύπτονται. Στο άρθρο 13 θα πρέπει να επεκταθούν οι υποχρεώσει διαφάνεια με τι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τι υποχρεώσει υποβολή πληροφοριών για τι εμπορικέ του συναλλαγέ. Επίση, εκτιμούμε την πρότασή σα να υπάρχει μια μέθοδο για τα κουρέματα ε, να συνάδει με αυτούς τους κανόνες και τις ε, σχετικές συστάσεις που θα προκύψουν σύντομα από το ε, Συμβούλιο του Συστημικού Κινδύνου. Ε, θα πρέπει να δούμε επίσης την πρόταση από τις εξής σκοπιές. Να συμπεριλάβουμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την δυνατότητα ε, κεντρικής παρακολούθησης και τις, ε, απαιτήσει διαφάνεια. Επίση, να προσθεθεί ένα άρθρο ώστε η ΕΣΜΑ να παρέχει ε, συγκεκριμένου κανόνε και πληροφορίε για του όγκου και το, τα στοιχεία των αντισυμβαλωμένων σε αυτή τη χρηματοδότηση, τη συναλλαγή χρηματοδότηση τίτλων. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει μια συνάθρηση των στοιχείων βάσει των ε, τεστ κοπόσεως που έγιναν ήδη και για την ε, ανταλλαγή τέτοιων ε, χρηματοδοτήσεων. Επίσης ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει τους νόμους αφαιραγγιότητας και την δυνατότητα τα STF να συνδυαστούν εδώ με αυτούς τους κανόνες, με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων και θα πρέπει να διακριθούν οι συμφωνίες επαναγοράς από τις ανταλλαγές εξασφαλίσεων, ώστε τα, τα ρέπος δηλαδή από τα collateral swaps και να είμαστε βέβαιοι για την αντοχή τους ε, σε χρηματιστηριακές ε, καταρρεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει όλη την προσοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να έχουμε υπόψη το λίγο χρόνο που μας απομένει. Ωστόσο θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος ο οποίος θα ήθελε να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία κατσουδιά για να κάνει κάποια ερώτηση. Βλέπω πως όχι, οπότε θα δώσω τον λόγο στον Πάτρικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Το πρώτο σημείο κατά πώ θα πρέπει οι μεταφορέ τίτλο να εξαιρεθούν του πεδίου εφαρμογή του κανονισμού. Τέσσερι λόγοι μα κάνουν να πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα ήταν καλή ιδέα. Πρώτον, με μια τέτοια εξαίρεση αυξάνονται οι κίνδυνοι. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μεταφορά ε, τίτλων και ανταλλαγής εξασφαλίσεων δεν υπάρχει καμία διαφορά, ούτε και ο κίνδυνος μειώνεται. Το θέμα είναι ο χρόνος, όταν αλλάζει δηλαδή η διοκτησία, η εξασφάλιση, αλλά και τα δύο, και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει ο παρέχοντα εξασφάλιση να λάβει πίσω την εξασφάλιση. Άρα ο κίνδυνο είναι ο ίδιο. Πρέπει να επιστραφεί η εξασφάλιση. Αυξάνεται και η ανασφάλεια δικαίου, λέει ο κλάδο, ότι αν δεν εξαιρούνται οι συναλλαγέ χρηματοδότηση τίτλων, αυξάνεται η ανασφάλεια δικαίου. Με την εξαίρεση συγκεκριμένα, αυξάνεται η ανασφάλεια δικαίου. Υπάρχει συγκεκριμένη απέτηση, αλλά αν αποκλείσουμε αυτό το μέσο, δίνουμε τη λάθος εντύπωση, ενώ υπάρχει συνένεση ότι δεν υπάρχει. Επίσης, αν εξαιρέσουμε τις αυγές χρηματώσεις τίτλων, το 95 με 6% της αγοράς εξαιρείται από την πρόταση. Αυτά τα λέει ο ίδιος ο κλάδος. Άρα υπονομεύουμε την πρόταση. Τέλος. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αν συμπεριλάβουμε αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει ο κλάδος πολύ απλά να αλλάξει τα γενικά πρότυπα και κείμενα. Να προσθέσει δύο-τρεις προτασούλες που να λένε ότι έχει δώσει συνένεση, παρέχουν την εξασφάλιση της αλλαγής χρηματοδότησης τίτλων. Συμφωνούμε απόλυτα με τον εισηγητή λοιπόν ότι είναι πολύ κακό να ε, εξαιρεθούν οι τίτλοι. Τώρα, δύο-τρία τελευταία σχόλια. Φυσικά και πρέπει να βρούμε τη λύση. Δεν μπορεί να απαλλάσσονται ή να είναι εκτό πρόταση κεντρικέ τράπεζε. Πάλι δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι οι κεντρικέ τράπεζε, στις αρχέ τη αγορά. Αυτό θα ήταν ένα πολύ κακό μήνυμα αν δεν μπορούσαν να δίνουν ε, στι δημοσιε αρχέ αγορά, πληροφορίε κεντρικέ τράπεζε και οι αρχέ δεν θα είχαν κανένα ρόλο μέσα σε αυτή την πρόταση, αφού δεν θα μπορούσαν να υποπτεύουν ε, να παρακολουθούν την εφαρμογή του κανονισμού. Ε, Απαιτήσει σε υποβολή εκθέσεων ναι, είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να μειώσουμε την, ε, το φόρτο εργασία. Επίση, θα πρέπει η υποβολή εκθέσεων να, να βασίζεται στου κανόνε που υπάρχουν. Γιατί με το position data θα έχουμε τι λάθος πληροφορίε Με το transaction reporting ουσιαστικά βασιζόμαστε στο ΕΜΗΡ και στα νύφη τους κανονισμούς που υπάρχουν. Άρα αυτός είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπο να προχωρήσουμε. Σε ό,τι αυτά τα κουρέματα, η καλύτερη ρυθμιστική προσέγγιση είναι. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος, ούτε το κόστος ε, για τον ε, κλάδο. Και αφού δεν γνωρίζουμε τι θα κοστίσει και τι αντίκτυπο θα έχει η ρύθμιση, ίσως το καλύτερο θα ήταν να ακολουθήσουμε τη συμβαστική πρόταση που ζητά μελέτη αντικτύπου, υποβολή έκθεση και εισαγωγή των κανόνων αφού υπάρξει διεθνή συμφωνία. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Ευχαριστώ. Thank you to the Commission. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα το λόγο έχει ο εισηγητή Ρενάτο, παρακαλώ. I thank you all for uh, your comments and for uh, your... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και για τα σχόλιά σας όλους. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα. Γιατί νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχουμε βρει συμβιβαστικές λύσεις σε πολλά θέματα. Compromise on the, in order to reduce the duties for the SMEs ε, συμφωνώ με αυτό που είπε η συνάδελφος Δανούτα Χούμπνερ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, η συμβιβαστική πρόταση όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό σημείο ε, επί του οποίου να βασιστεί η συζήτηση για τη συμβιβαστική λύση. Άκουσα τις αιτιολογήσεις των άλλων σκιωδών εισηγητών και τις επεξηγήσεις τους όσον αφορά την δυνατότητα αποφυγής της εφαρμογής ε, του κανονισμού για την συλλογική συμφωνία μεταφοράς ε, τίτλων, έτσι όπως την ονομάζουμε. Πιστεύω ότι αυτή η εξαίρεση θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για την ε, έκθεση, γιατί αυτομάτως βγάζουμε απ' έξω το 25% των συναλλαγών και της αγοράς. Η διαφάνεια βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική και ήταν μάλιστα ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία μας. Και το σημαντικό είναι να, ε, να δούμε το σημείο αυτό σαν ε, τμήμα της διορθωτικής αλλαγής ε, της αγοράς τίτλων και της τραπεζικής αγοράς, έτσι ώστε να αποφευθούν στο μέλλον συστημικοί κίνδυνοι. Πιστεύω ότι αν θέλουμε πραγματικά να αποφύγουμε τους συστημικούς κινδύνους θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η αγορά σήμερα ε, και να ε, καταλάβουμε ότι αν δεν θέλουμε προβλήματα στο μέλλον θα πρέπει να ρυθμίσουμε καλύτερα την αγορά. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε επιτύχει μια πολύ καλή βάση ε, επί της οποίας μπορούν να στηριχτούν συμβιβασμοί. Στις επόμενες ε, ημέρες θα συνεργαστούμε έτσι ώστε να εξευρεθούν περαιτέρω συμβιβασμοί επί μεγαλύτερου τμήματος της προτάσεως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή, ευχαριστούμε τους σκιώδεις. 23 Μαρτίου θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση με το θέμα αυτό. Είναι, να μην το λησμονούμε αυτό, ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Τώρα έχουμε το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, στο οποίο μπορούμε να περάσουμε άμεσα. Είναι άμεσα συνδεδεμένο μάλιστα, γιατί αφορά τα διορθωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστοτικών ιδρυμάτων. Έχουμε πολλέ τροπολογίε, ήταν εύκολο να το ε, σκεφτείτε αυτό και να το καταλάβετε. Τώρα για να τα μελετήσουμε όλα αυτά τα σημαντικά και ενδιαφέροντα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Χόκμαρ Γκούναρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους Σκιώδης και τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει όλε αυτέ τι τροπολογίε. Δεν θα έλεγα ότι είναι λίγε. Από την άλλη, ευτυχώ επικεντρώνονται στα βασικά ζητήματα. Υπ' αυτήν την έννοια, λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι είναι απλά τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον είναι εφικτό να βρούμε ε, έναν τρόπο να το οργανώσουμε σε κατηγορίες και σε ομάδες για να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ήθελα να τονίσω με κάποια σύντομα σχόλια Πρώτα απ' όλα, τροπολογίες για το είδος αυτός εμπορίας και για το τι είναι η δημιουργία αγοράς και πώς μπορεί να έχουμε εναλλακτικά προϊόντα. Αυτά είναι δύο ζητήματα που θα μας επιτρέψουν αν τα λύσουμε να έχουμε νομική ασφάλεια. Είναι εφικτό να βρεθεί ευολύση. Αλλά ίσως χρειάζονται περισσότερες, ενώ υπάρχουν μάλλον τόσες απόψεις για την τράπεζα, για το property trading και το market making, όπως λέγονται, ε, υπάρχουν τόσες απόψεις όσο και για την ψηφιακή όχι διάσταση των τραπεζών. Είναι σημαντικά αυτά ε, μεταξύ μας ε, να τα λύσουμε και υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες από τις συζητήσεις που είχαμε και γι' αυτό θα επικεντρωθώ στις διαφορετικές τροπολογίες ε, για τις επιδοτήσεις. Ε, και εγώ είχα την άποψη ότι θα πρέπει να, με, την τράπεζα, με την οδηγία για την τράπεζα το, της των, με την οδηγία για την εξηγία των τραπεζών να έχουμε απειλήσει αυτό το ζήτημα. να δούμε αυτές τις έμεσες επιδοτήσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η μεταρρύθμιση της δόμη των τραπεζών, αλλά και τι μήνυμα θα δώσουμε στον τραπεζικό κλάδο και την όλη κοινωνία. Εκεί δεν θα πρέπει και θα πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει καμία έμεση έμεση επιδότηση προ οποιοδήποτε ε, μέτοχο. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν οι μέτοχοι ότι δεν θα υποφεληθούν από κανένα μέτρο διάσωση, είτε από το Ταμείο για την Εξυγένση, είτε από τι κυβερνήσει. Αυτό ήταν από τα μεγάλα ζητήματα που μα απασχόλησαν ε, την οδηγία για την εξηγήση των τραπεζών. Και εδώ είναι σημαντικό αυτό να δηλωθεί ευθύ εξ αρχή. Είναι σαφέ ότι όσοι είναι senior ε, επενδυτέ, Πρέ, προφανώς ασχολούνται με το γεγονός του αν θα υπάρχει διάσωση με ίδια μέσα γιατί είναι πιο εκτεθειμένοι. Αλλά εφόσον υπάρξει παρέμβαση, ε, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε ότι όχι δεν θα υπάρξει παρέμβαση, αλλά ως προς τις θέσεις συνέχεια θα μας απασχολεί το πώς πρέπει να καλύψουμε τους καταθέτες για καλούς κακούς λόγους, για πολιτικούς ή όχι λόγους, για μια σειρά από λόγους. Αλλά Νομίζω είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι εν μέρει αυτό το λύσαμε με το σύστημα αγγίσεως των καταθέσεων. Κύριε Σάιμον, θα ήθελα να είστε στο πλευρό μου. Και νομίζω ότι έχουμε προβλέψει εδώ κάποια νομική κάλυψη. Όμως είναι ενδιαφέρον διότι ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα σε αυτή την Επιτροπή όπου ε, καταλήγουμε να θέλουμε να δώσουμε έμεση επιδότηση προς το τραπεζικό σύστημα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ουσιαστικά έμεση επιδότηση είναι αυτό. Και ήθελα να το πω, να το δηλώσω. Το παράδοξο εδώ είναι ότι αυτές οι έμεσες επιδοτήσεις ουσιαστικά θα υποφελήσουν τις τράπεζες. Ενώ οι επιδοτήσεις που είναι ε, πηγαίνουν υποτίθεται στην πραγματική οικονομία και εκεί που έχει χαμηλότερα επιτόκια. Αυτά όλα λοιπόν είναι πράγματα που συμβαίνουν και προκύπτουν πολλέ απορίε. Νομίζω όμω ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Είμαι σχεδόν σίγουρο και για μένα ήταν πολύ σημαντικό να συσχετίσουμε την μεταρρύθμιση τη δομή των τραπεζών με την οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Διότι όσο πιο πολύ ε, συσχετιστούν, τόσο πιο αξιόπιστοι θα είμαστε με την ε, οδηγία για την εξυγίαση των τραπεζών και την όλη αυτή διαδικασία του Μπέιλιν, τη της διάσωσης με ίδια μέσα. Κάτι άλλο που ανέκυψε στις συζητήσεις και που αφορά κυρίως τις τροπολογίες που είναι οι χώρες ε, προέλευσης και οι χώρες υποδοχής. Ε, ο κύριος Κάριν και ο κύριος Ροζάτη ε, θέλουν να δούμε ακριβώ τι ισορροπία θα βρούμε μεταξύ του home και host, δηλαδή τη χώρα ε, προέλευση και τη χώρα υποδοχή. Εάν αυτό δεν καλυφθεί εδώ, υπάρχει περίπτωση οι χώρε αυτέ που έχουν ε, κατεξοχήν τράπεζε ε, ξένες, ξένης προέλευση και εφόσον γίνει διαχωρισμό. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι ευρέω είναι περίπου αποδεκτή. Θα υπάρχει συρρήκνωση τη ε, εξασφάλιση ύπαρξη τιμών αγορά και πώληση ε, στις χώρες αυτές, σε χώρες όπως η Λετωνία, η Λιθουανία και η Εστονία, ε, η δική τους η δική τους η πλευρά της αγοράς, του market making όπως λέγεται, εξαρτάται πολύ από άλλες χώρες. Αυτή η λειτουργία λοιπόν θα περάσει ουσιαστικά, εάν υπάρξει συρρήκνωση, στις χώρες αυτές όπου βρίσκονται και τα κεντρικά της τράπεζας και τα βασικά κεφάλαια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε για πολλούς ε, σοβαρούς λόγους και για την Τραπεζική Ένωση, αλλά γιατί υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ότι το τόνισαν πολλοί συνάδελφοι. Η ανάγκη δηλαδή διευκόλυνσης των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τώρα αναλάβουμε μέτρα που δυσκολέψουμε την, ε, με την κίνηση των κεφαλαίων, τις συναλλαγές και τη δανειοδότηση, αυτό θα επηρεάσει όχι μόνο τις χώρες ε, υποδοχής, αλλά και τις χώρες προέλευσης στην οικονομία τους. Έχουν γίνει πολλές συζητήσει για τον αν θα έχουμε μια προσέγγιση διαρθρωτικού τύπου ή βάση του κινδύνου. Νομίζω μια τάση των... που διαφαίνεται από πολλές τροπολογίες είναι πώς να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους. Και αρκετές τροπολογίες υπογραμμίζουν το γεγονός ότι συστημικοί κίνδυνοι εντοπίζονται και πολλές φορές προέρχονται από μικρές τράπεζε, όχι μόνο από μεγάλες. Αυτό έχει να κάνει με την ε, περιπλοκότητα του σύγχρονου τραπεζικού συστήματο, όπου μεγάλε και μικρέ, γενικώ οι τράπεζε, είναι αλληλεσχετιζόμενε τόσο πολύ, αλληλένδετε, που ε, αν το λέγαμε φιλοσοφικά, θα λέγαμε ότι κάθε τράπεζα είναι υποκατάστημα μια άλλη ε, μεγαλύτερη στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα. Αυτό έγινε με του αδερφού Λίμαν με μια πολύ εξειδικευμένη τράπεζα επενδυτικών προϊόντων που όμως είχε και συστημικό αντίκτυπο από ό,τι φάνηκε στο όλο τραπεζικό σύστημα. Πολλές είναι λοιπόν οι τροπολογίες που τονίζουν την ανάγκη να επικεντρωθούμε στην ε, εξηγενσιμότητα. Εάν σκεφτούμε τι συζητήθηκε ως τώρα και οι τροπολογίες έχουν υποβληθεί, φαίνεται να υπάρχει αυτή η διαφορά στις προσεγγίσεις. Ή συστημικός κίνδυνος ή εξασφάλιση της δυνατότητας εξυγίευσης. Για μένα, η εξασφάλιση της, εξυγεία, της δυνατότητας εξυγίευσης είναι ο τρόπος να μειώσουμε τους συστημικούς κινδύνους. Αυτή είναι η εξασφαλιση της δυνατοτητας εξυγιανση για μενα η εξασφαλιση της της δυνατοτητας εξυγιευσης προσέγγιση. Και υπ' αυτήν την έννοια, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αν δω όλες τις τροπολογίες. Τι βλέπω ο κ. Φαντάιζε και είπε την περασμένη φορά ότι απέχουμε πολύ μεταξύ μα, ότι από την πλευρά του έρχονται παγωμένοι άνεμοι. Δεν το πιστεύω αυτό. Εάν, δεν το πιστεύω εγώ αυτό, γιατί εάν μπορέσουμε να εντοπίσουμε πού είναι οι διαφωνίες μας σε συγκεκριμένα σημεία και να μην μείνουμε στα συμβολικά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί και εγώ θέλω να έχουμε ένα ευρωστότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τον συστημικό κίνδυνο και τα προβλήματα που προκύπτουν. Δεν υπάρχει κανείς, ακόμη κι αν κάποιες φορές στα λόγια μα ε, φαίνεται κάτι αντίθετο. Κανεί δεν υποτιμά την ανάγκη να έχουμε περισσότερε επενδύσει. Και κανεί δεν λέει ότι οι χώρε υποδοχή δεν θα πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα του market making, της εξασφάλισης ύπαρξης τιμών αγοράς και πώλησης. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν αυτήν την ανάγκη market making και για μένα έχει ανοίξει ένας δρόμος ε, δυνατότητας εξέβρεσης συμβασμών. Το προσπαθήσαμε να μην μακρηγορήσω πρόεδρε. Ε, να αντιμετωπίσουμε τις συγκεκριμένες μας ε, δυσκολίες και διαφωνίες και όχι τα θεωρητικά. Δηλαδή, υποχρεωτικός διαχωρισμός ή όχι. Εάν μείνουμε σε θεωρητικές τέτοιες διαφιλονικίες θα έχουμε πολύ μεγάλες διαφωνίες. Αλλά νομίζω ότι του συγκεκριμένου, οι τράπεζες που έχουν ένα τεράστιο μέρος της αγοράς στα χέρια τους, αλλά με πολλές διακυμάνσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καλύψουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ή τέλο πάντων να λύσουμε το πρόβλημα ότι κάποιε μεγαλύτερε τράπεζε μόνο και λόγω του μεγέθου του μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα από τι μικρότερε και αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα των ε, χωρών ε, υποδοχή και προέλευση και αυτό νομίζω ότι μπορεί να επιληθεί. Νομίζω, Πρόεδρε, και τώρα σα απευθύνομαι ω εκπρόσωπος του υπέροχου και μεγαλειώδους έθνους της Ιταλίας που είστε, ε, να θυμίσω ότι στην Ιταλία εφευρέθηκε η σύγχρονη οικονομία από τις αρχές της Ιταλικής λογιστικής. Ε, εάν δεν έχω παραπληροφορηθεί, πολύ κοντά στην πόλη του Γκουαλτιέρη, κοντά στη Γένοβα ή στη Βενετία, στις ε, θαλάσσιες αυτές δημοκρατίες, όπου η λογιστική καταγραφή των τραπεζικών στοιχείων δείχνει τη διάσταση της νοοτροπίας που υπήρχε και την πολιτιστική αξία. Αλλά σκεφτείτε όλοι όσοι περάσατε και από τις συμπληγάδες του double account, accounting στις σχολές σας ή στα πανεπιστήμια σας. Ε, ο συσχετισμός πολλές φορές έχει να κάνει με το πόσο συνδέουμε την πραγματική οικονομία με τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό ήταν ο στόχος του double accounting, της διπλής λογιστικής των διπλών λογιστικών υπολογισμών. Αυτό λοιπόν είναι η προοπτική μας. Εάν δούμε όλες τις τροπολογίες, ε, εάν δούμε όλες τις τροπολογίες, σκεφτόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ένα νέο επίπεδο διαφάνειας. Θα μπορούσα να το ονομάσω αυτό ε, βενετσιάνικο παράθυρο. Με τη λογική ότι από τη μια άποψη έχουμε αγορά και εμπορευομένους, αλλά με επόπτες που θα έχουν περισσότερα στη διάθεσή τους να δουν, να, παρακολουθήσουν και να αναλύσουν. Και η διαφάνεια θα υποχρεώσει τις αρχές να δράσουν όταν είμαστε υποχρεωμένοι να δράσουμε. Δεν θα κρύβονται πια, δεν θα, είναι, δεν θα κουκουλώνονται τα προβλήματα. Αλλά το θέμα αυτό πρέπει να διασυνδεθεί με την ίδια την αγορά, διότι όταν συζητούμε την οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα είναι ότι όποτε ένας επενδυτή χρειάζεται να βεβαιωθεί την επένδυσή του, δεν πηγαίνει σε πολύ επικίνδυνες κατευθύνσει, τότε κινητοποιούνται πολλοί από τους επόπτες του επιχειρηματικού κόσμου, του τραπεζικού κλάδου. Είναι λοιπόν ένα θέμα που μπορεί να λυθεί εάν στο επιχειρηματικό κομμάτι των εμπορικών συναλλαγών υπάρξει περισσότερη διαφάνεια. Εκεί θα δούμε και τα μοτίβα που ακολουθούν ε, οι διάφορε συναλλαγέ, τι διακυμάνσει του. Την ε, περίπτωση να ανοίξουν αυτά τα βενετσιάνικα παράθυρα και να δράσουν οι αρχές. Όχι μόνο με τον υποχρεωτικό διαχωρισμό, αλλά ε, και άλλα εργαλεία ώστε οι αρμόδιες αρχές να δράσουν, όχι μόνο βάσει των δικών τους απομονωμένων γνώσεων, αλλά βάσει της ε, ευρύτερης γνώσης. Έτσι θα ενισχύσουμε το εύρος των, του συστήματος συνολικά. Όχι υποχρεώνοντας ε, τις επενδύσεις ή τις χρηματαγορές σε σκιώδεις ε, περιοχές του ταπεζικού συστήματος, αλλά με περισσότερους κανόνες και με ένα πολύ σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο αντιμετώπιση του όλου συστήματο. Έτσι ε, αντιλαμβάνομαι τι νοοτροπίε, τι ε, τις τροπολογίες και έτσι νομίζω μπορούμε να βρούμε εφικτέ συμβαστικέ λύσει. Πρόεδρο. ευχαριστούμε τον εισηγητή. Καλωσορίζουμε την αισιοδοξία σα για, για αυτό το δρόμο που ανοίγεται για συμβαστικέ λύσει. Έχουμε και τι ευλογίε ε, του Λούκα Πατσόλη και ότι χρειάζεται για, τις, ε, για τα διπλή καταγραφή στοιχείων αλλά να μην ξεχνάμε και τα 8 δι από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Είναι αρκετά για τι επιδοτήσει προ τι τράπεζε. Πολύ ωραία θα ήταν να ίσχυε αυτό, αλλά δεν συμβαίνει. Τώρα να, να ακούσουμε τα σχόλια του εισηγητή των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον Κούναρ για αυτή την εξαιρετική εισαγωγή του. Ε, μακάρι να μπορούσα να συμμεριζόμουν κι εγώ αυτό, αυτή την αισιοδοξία σας. Και πραγματικά θα ήμουν περιχαρής αν μπορούσατε να δεχτείτε κάποιες από αυτές τις 700, πάνω από 700 τροπολογίες. Δυστυχώς όμως πίστευα πως ε, βρισκόμαστε ακόμα στα βασικά, στα πρώτα στάδια της ανάλυσης του τι συμβαίνει και η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι πολύ, αυτά πολύ μεγάλα ιδρύματα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση από τον Charles Goodhart σε μια από τις ακροάσεις που κάναμε, κατά την οποία ανέφερε την έννοια του Μπέιλιν, in αυτής της διάσωσης με τα ίδια μέσα και πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσει καλά σε μια συστημική κρίση. Επίσης είχαμε και την πράσινη βίβλο για την Ένωση των Κεφαλαίων και θα ήθελα να σας διαβάσω ένα κομμάτι από αυτήν που καθιστά σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, τις, ε, έχει παρόμοιες απόψεις. Μιλάει λοιπόν για την αύξηση των κεφαλαίων τις τελευταίες δύο δεκαετίες η οποία σχετίζεται άμεσα με την ανταλλαγή χρεών και τα ομόλογα αγοράζονται από χρηματοπιστωτικές ε, εταιρείες, πολλούνται από άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες, αλλά αντί να έχουν όφελος για τον τελικό καταναλωτή και να αυξάνουν την ε, διαλειτουργικότητα, αυξάνουν τους συστημικούς κινδύνους. Ε, ταυτόχρονα Μόνο ένα πολύ μικρό ε, μέρος των εμερισμάτων αφορά μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες ως ε, αντισυμβαλόμενους και πιστεύω πως αυτό καθιστά σαφές ότι εάν συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα επίπεδα ε, διασυνδεσιμότητας θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε too big to fail πολύ μεγάλα ζητήματα, πολύ μεγάλα ζητήματα για να τα αφήσουμε να καταρρεύσουν. Πιστεύω πως εδώ δεν είμαστε μόνο στη θεωρία, αλλά σκεφτόμαστε και πρακτικά και βλέπω μία διαφορά ανάμεσα στην βασική ανάλυση που έχει γίνει εδώ. Δεν είναι ανήκουστο να βρίσκονται συμβιβασμοί όταν υπάρχουν διαφορές, θεμελιώδεις διαφορές στην ανάλυση. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι θεμελιώδεις διαφορές και ότι δεν είναι στη σφαίρα της θεωρίας. Τώρα, όσον αφορά το που οδεύουμε, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την πρόταση Μπαρνιέ ε, ως έναν πάρα πολύ καλό συμβιβασμό ανά, μέσα στην ε, προσέγγιση του Βίκα που ήθελε να διαχωριστεί η λιανική τραπεζική από, τη, από τις τράπεζες και που προέβλεπε ένα, μια απαγόρευση στην, ε, στο εμπόριο αυτών των αξιών. Ο στόχος λοιπόν της αρχικής πρότασης Μπαρνιέ είχε ως εξή. Πρέπει να πάρουμε τα πλεονεκτήματα του Ευρωπαϊκού Γενικού ε, Καθολικού Τραπεζικού Συστήματος, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτήν την Καθολική Γενική Τραπεζική να συνεχίσει ως έχει. Δεν είναι θέμα λοιπόν μεγέθους, είναι θέμα του τι κάνουμε με αυτό το μέγεθος. κινούμαστε στα περιθώρια ή εντός ορίων. Αυτή λοιπόν η απόφαση δεν είναι μια απόφαση που, την οποία μπορούμε να πάρουμε λέγοντας ναι ή όχι, είναι, ε, έχει διαβαθμίσεις. Και πιστεύω πως ήδη έχει αναφερθεί σε αυτή την Επιτροπή, αλλά αξίζει πιστεύω να το αναφέρω άλλη μια φορά. Υπάρχουν αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αρκετά μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν κάτω από 40% κεφαλικές ε, συναλλαγές. Όμως, αυτό λοιπόν είναι ένα μόνο μέρος των εργασιών τους. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό μοντέλο όσα έχει λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τις γενικές τραπεζικές εργασίες. Τώρα κάτι άλλο. Τι γίνεται στην πράξη. Και είμαστε όλοι πρακτικοί άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ πώς μπορούμε να κάνουμε σωστά αυτήν την ε, τραπεζική εποπτεία στην πράξη. Η απάντηση είναι πολύ σύντομη. Ότι ακόμα και σήμερα ο ΙΣΕΣΕΜ έχει τη δυνατότητα εφόσον θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος να επιβάλλει διαφοροποίηση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Γι' αυτό λοιπόν, εάν εσεί πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη ε, χεμήθεια και ότι δεν υπάρχει ε, κάποιο πρόβλημα που είναι υπερβολικά μεγάλο για να το αφήσουμε να αποτύχει, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Όμως, αν θέλετε απόλυτη χεμήθεια, έχετε τη δυνατότητα να επιβάλλετε αυτές τις, τις διαφοροποιήσεις. Όμως είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του, γιατί φανταστείτε, είστε εσεί ένα από αυτού του επόπτε και έχετε αυτή την ε, θεωρητική εξουσία να το κάνετε αυτό. Όμως στην πράξη, όταν αντιμετωπίζετε μία άμεση χρηματοπιστωτική κρίση, θα ε, καταλήξετε να ακολουθήσετε τη δικαστική οδό, θα πάτε στα δικαστήρια και τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται λοιπόν ε, να υπάρχουν όρια, χρειάζεται να υπάρχουν λοιπόν ε, να υπάρχει ε, αυτό το βάρος των ε, αποδείξεων σε αυτά τα όρια το μη αναστρέψιμο βάρος των αποδείξεων και γι' αυτό πιστεύω πως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα και να επιστρέψουμε στην αρχική πρόταση Λικάν με, για ένα δεύτερο όριο, ένα δεύτερο κατόφλι, όπου αυτός ο διαχωρισμός δεν θα είναι πλέον στη δυνατότητα και στη διακριτική ευχέρεια του επόπτη, αλλά θα γίνεται αυτόματα. Και πιστεύω πως ε, έτσι μπορούμε να πλησιάσουμε λίγο τα όσα συζητούνται στο Συμβούλιο και ε, να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο του φαναριού, του φωτεινού σηματοδότη. και να, συνδυά, και να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα φωτεινό σηματοδότη όπου ακόμα και αν δείχνει κόκκινο να υπάρχει η δυνατότητα για διαφοροποίηση, για αλλαγή πορείας. Και πιστεύω πως και αυτό είναι το νόημα των τριών χρωμάτων, έτσι, σε αυτό το φωτεινό σηματοδότη, που πιστεύω πως είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Ε, τώρα, θα ήθελα να αναφέρω και μια άλλη τροπολογία, η οποία έχει να κάνει με αυτό το πρόβλημα. συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό. Θα ήθελα να δοθεί περισσότερη έμφαση στην απαγόρευση αυτών των συναλλαγών και να δούμε πώς μπορούμε να μοχλεύσουμε ένα αλλακτικό ε, ταμείο επενδύσεων. Διότι στα πλαίσια της ε, Ένωσης Κεφαλαιαγορών πρέπει να προσέξουμε να μην οφήσουμε όλες αυτές ε, τις ε, συναλλαγές στην, ε, στις στο σκιώδη τραπεζικό χώρο. Και γι' αυτό εμείς προτείνουμε να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα, να γίνει πιο αυστηρή η αρχική πρόταση. Και βλέπω πως μου τελειώνει ο χρόνος, Πρόεδρε, γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω και ένα ε, τρίτο σημείο, το τι γίνεται δηλαδή και πώς, ε, πώς μπορεί να υπάρξει λειτουργία κάτω από ε, πολλαπλές δικαιοδοσίες όπως και οι πάρα πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται υπό έλεγχο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και πέρα από αυτό και πώς θα το συνδυάσουμε αυτό με τον έλεγχο αμερικανικών τραπεζών. Πρέπει να δούμε πώς αυτή η μία θηρίδα επίλυσης από θεωρία θα περάσει στην πράξη. Και όταν μιλάμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πιστεύω πως δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στο βίκαρι βόλκα στο ποια μέθοδο θα ακολουθήσουμε, αλλά σε αυτή τη, σε μία εξυγίανση, όχι με μία μόνο θηρίδα, αλλά πολλαπλές και υπάρχουν τροπολογίες που έχω υποβάλει σχετικά. Θα σταματήσω όμως εδώ και δεν θα επεκταθώ, αλλά στην πορεία με τα χαρά να σας το αναλύσω. Ευχαριστώ πολύ για την ίσια ο Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε μήπως ε, μπορέσω να συνεισφέρω στην ε, προσέγγιση των δύο ομάδων. Η ε, ειρήνη, η αγάπη ο Τζίμι Χέντριξ άλλωστε ήταν ο αγαπημένος μου τραγουδιστής ε, που γράφει σε ένα τραγούδι του ότι οι σηματοδότες αύριο θα γίνουν μπλε. Άρα πρέπει να ξέρουμε με αυτούς τους σηματοδότες τι καλύπτουμε. Να προετοιμαστούμε, όπως ε, λέει και το έργο μας στο Μαύρο Κίκ, για το απροσδόκητο. Ας περάσουμε λοιπόν ε, στην ουσία. αν δεν κανείς τροπολογίε άλλων και τι δικές μου. Πιστεύω ότι όπως και άλλοι, και εγώ εκείνο βέβαια από την αρχή, ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε στις τράπεζες να καταρρεύσουν. Δεν μου αρέσει όμως να πληρώνουν για τη διάσωσή τους οι φορολογούμενοι. Σε, αυτό, σε αυτή την πρόταση, σε αυτό το σχέδιο έκθεσης, συμφωνούμε νομίζω όλοι μάλλον παρακάπνισα, δεν μπορώ να εκφραστώ καλά, τη διασταύρωση των επιδοτήσεων. Δεν θέλουμε να στρεβλώσουμε όμως την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο λοιπόν το ε, το, όσο το περισσότερο, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν κρατικές επιδοτήσεις και ούτε φαλούμε να πληρώνουν για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν κάποιοι. Υπάρχουν και τροπολογίες του κυρίου Λάμπερτς και του κυρίου Ντεμάση, του Φανβάι Ζέκερ που πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Άρα συμμερίζονται και άλλες πολιτικέ ομάδες πιστεύω την άποψή μα. Σε ό,τι αφορά πιστοτικά ιδρύματα μέτρα τρίτες χώρες το έθεξαν και άλλοι παρουσάρι στη Σιγκαπούρη στις ΗΠΑ. Άρα αυτά τα πιστοτικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογή κανονισμού για να μην πιάνονται εισαγωγικών δύο φορέ. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο κανονισμό αυτό τις ε, συνεταιρισμού του τραπεζικού ή τις ασφαλιστικές εταιρείε να μην τις περιλαμβάνει. Θα ήθελα να δούμε και ποιες αριθμητικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται. Σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, το prop trading, απαγόρευση του prop trading. Η λέξη position που χρησιμοποιείται συνήθως έχει να κάνει με μέσα και με συναλλαγές, άρα δεν θα συμφωνούσα. Entry into νομίζω είναι καλύτερη λέξη, καλύτερο, καλύτερη έκφραση. Τα τελευταία πέντε χρόνια που ήμουν στην Επιτροπή και αν σκεφτώ τι συζητήσαμε με το EIFMD νομίζω ότι την αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου την ψηλοκαταστρέψαμε όπως και πολλά άλλα. Οπότε λέμε ας βρούμε μια λύση. Α, ναι, ο ECF είναι η λύση. Εμείς δεχόμαστε να ρυθμίζεται η κίνηση κεφαλαίων με αυτό το μηχανισμό. αλλά μπορεί να μην θέλουμε στο ταμείο αυτό να συμμετέχουν οι τράπεζες. Υπάρχουν και επενδυτές όμως, ε, ιδιώτες, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση και ξέρουν τα αποθέματα που έχουν μεγάλα πιστοτικά ιδρύματα. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους αποταμιευτές. Γι' αυτό και εγώ βάζω τη λεγόμενη qualifying deposit ως ορισμό. Επίσης θεωρώ και δεν το Βρετανός Εάν κάθε κράτος μέλος έχει ένα σύστημα που αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, εμείς πρέπει να προσέξουμε να μην υπονομεύσουμε τις εθνικές λύσεις. Συνάδελφοι άλλων χωρών έχουν έρθει και μου έχουν πει ότι δεν τους πείραζε η οδηγία να ήταν η αντίστοιχη ρύθμιση Vickers που να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ όμως λέω ότι πρέπει να εφαρμόζονται τα σωστά μέτρα αναζητούμε ίσως ένα μέγεθος ε, κοινό για όλους. Αλλά δεν θα έπρεπε να υπονομεύσουμε εθνικέ λύσεις που μπορούν να λειτουργούν. Θα καταθέσω λοιπόν τροπολογίες. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ευελιξία. Και το σύστημα να είναι εύρωστο. Ιδίω για όσε χώρε έχουν προχωρήσει τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα υποδοχή, home host, το κάλυψαν προλαλήσαντε συνάδελφοι, δεν θέλω να εξέλθω λοιπόν σε λεπτομέρειε. Τρει-τέσσερι είναι οι τομεί όπου εγώ θα καταθέσω τροπολογίε. Σα τι προανέφερα. Η ομάδα μου συνολικά, πρέπει να σα πω, στηρίζει την προσέγγιση Hackmark. σω να είμαι εγώ λίγο πιο ριζοσπαστικό σε σχέση με άλλα μέλη τη ομάδα μου. Οι αρχέ όμω ε, που είχα ήταν πάντα τρει. Να μην διασώζουν οι φορολογούμενε τράπεζε Δεύτερον, να αφήνουμε όπω συμβαίνει σε οποιοδήποτε άλλο τομέα και τι μεγάλε τράπεζε να καταρρεύσουν, γιατί είναι υπάρχει διαφορά εκεί και γιατί κάποιο να περιμένει να τον σώσει ο φορολογούμενο. Και πώ θα προετοιμαστούμε για την επόμενη κρίση, αν συμβεί. Το θέμα είναι οι διευθυντέ, το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι αυτό που θα αναλάβει την ευθύνη και να μην πληρώσουν φορολογούμενοι, αλλά να επιτρέψουμε να καταρρεύσει μια μεγάλη τράπεζα. Γιατί όχι. Ε. Sorry, sorry, Sylvie, sorry. Η Σιλβί, Σιλβί Γκουλάρ, ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο. Ένα μικρό λαθάκι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Κούναρ και όλου του άλλου εισηγητέ οι οποίοι καταβάλουν τεράστια προσπάθεια επί του θέματο αυτού. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε έναν τόπο κοινό. Ε, το είπε και ο Σαϊτ Καμάλ πριν από λίγο, αλλά και ο Γιάκο πριν, ότι συνειδητοποιούμε όλοι ότι υπάρχει η έννοια του κινδύνου και επομένως και της εποπτείας θέλουμε να, να διαγράψουμε τον κίνδυνο για τους φορολογούμενους, από την άλλη μεριά όμως να μπορούμε να παρεύουμε βεβαίως με τρόπο σαφώς καθορισμένο. Τώρα, εάν συμφωνήσουμε επί της αρχής, ο τρόπος παρέμβασης, αν θα έχουμε κατόφλι ή όχι, αν θα έχουμε φωτεινού σηματοδότηση ή όχι, θα το βρούμε αργότερα. Το πρώτο σημείο που το οποίο θα πρέπει να, να συμφωνήσουμε είναι εάν όλοι θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε ένα κίνδυνο κίνδυνο. Και όπως άλλωστε υπενόησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ε, γνωμοδότησή της, ε, τουλάχιστον για τις χώρες της Ευρωζώνης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε προσέγγιση η οποία να δίνει στον επόπτη περισσότερες ευθύνες, αρμοδιότητες. Ε, δεν θα συμφωνήσω με τον Γιάκο, ότι μπορεί να υπάρχει αυτοματοποίηση, ναι ή όχι, άσπρο ή μαύρο. Ε, θα πρέπει να δούμε και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά. Έχω την εντύπωση ότι και από αυτού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το δεύτερο σημείο επί του οποίου επέμεινε ο Γκούναρ στην έκθεσή του και νομίζω ότι είναι προσφυλές σε όλους μας είναι να βρεθεί καλή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία έναντι κινδύνου ε, και την δυνατότητα της μη χρηματοδότησης της οικονομίας, το ενδεχόμενο μη χρηματοδότηση της οικονομίας. Είναι πάρα πολύ, ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό ε, στην κοινή μας προσέγγιση να λάβουμε υπόψη μας την ανάγκη χρηματοδότησης της οικονομίας, ε, ε, την ανάγκη να έχουμε ανταγωνιστικό τραπεζικό τομέα, αλλά και την ανάγκη να εξακολουθήσει να είναι κυρίαρχος ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας. Αυτά θα πρέπει να σκεφτούμε, να φανταστούμε πού θα φτάσουμε εάν θα έχουμε ακόμα ευρωπαϊκές τράπεζες, θα μπορούσαν να είναι μέσα σε μια ενιαία δομή ή μοναδική δομή θα, θα πρέπει να δούμε στο τέλος της ε, διαπραγμάτευσης και της ε, συζήτησης εάν ε, θα υπάρξουν στο τέλος τράπεζες ευρωπαϊκές. Εγώ πιστεύω ότι οι τράπεζες παίζουν διαφορετικό ρόλο σε μια οικονομία από ότι ας πούμε μια εταιρεία η οποία κάνει παπούτσια ή παράγει iPhone. Η λειτουργία τους είναι διαφορετική, η λειτουργία των τραπεζών λέω, είναι διαφορετική από την μεταποιητική βιομηχανία, από τη βιομηχανία ή από τη γεωργία. Είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε αυτό και να συμφωνήσουμε από αυτού. Κάτι άλλο το οποίο μου είναι ιδιαίτερο προσφυλέ και αναφέρθηκε προηγουμένω είναι η ενιαία αντιμετώπιση τη τραπεζική αγορά. Πληρώνουμε υπερβολικά τον κατακαιρματισμό. Ε, οπισθοδρομήσαμε κατά τη διάρκεια τη ε, κρίση και ε, θα πρέπει τώρα μέσα από συγκεκριμένη νομοθεσία να ξεπεράσουμε αυτά τα βήματα προ τα πίσω. Το είπε και ο Γκούνερ, το είπε και άλλοι. Μερικές χώρε πήραν και μονομερή μέτρα και πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν πλέον να μην μπορέσουμε να φτάσουμε στη συμφωνία από αυτού του κειμένου, γιατί αν δεν επιτύχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες, τότε θα έχουμε κατακαιρματισμό, θα συνεχίσουν οι χώρες ε, οι οποίες έχουν ήδη πάρει μονομερή μέτρα να τα παίρνουν και επομένως θα σπάσουμε την αγορά, πράγμα το οποίο εγώ δεν θέλω ούτε καν να το φανταστώ. Πολύ σύντομα γιατί νομίζω ότι όλοι μακρηγόρησαν. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί κάποιων αρχών κατά την άποψή μου είναι ένα σύστημα risk-based, ε, συγκεκριμένες αρχές ε, για την ε, εποπτεία, όχι οπωσδήποτε τυφλή διακριτικότητα αλλά και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, αλλά μια σωστή τα επιβλεπόμενη κατάσταση, μία ρήτρα αναθεώρηση γιατί θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δούμε αργότερα τι θα κάνουμε, να ληφθούν υπόψη όλες οι πρόοδοι, θέλετε ή να το πούμε καλύτερα όλες οι αλλαγέ, οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε σχέση σε σχέση με, το, με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Το συγκεκριμένο τρόπο θα τον δούμε και ευελπιστώ ότι θα ακολουθήσουμε την οδό την οποία έχει καταδείξει ήδη ο εισηγητής και που γνωρίζω ότι ακολουθούν ορισμένες πολιτικές ομάδες, δηλαδή οδό προόδου δεν νομίζω και το λέω και το ξαναλέω ότι μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας μια αποτυχία που θα σημαίνει ότι η Κομισιόν θα αποφασίσει στη θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ Σιλβί, λέει ο Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη γιατί έκανα λάθος. Τώρα όμως θα δώσω το λόγο στην Κουεφάβιο Δεμάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάθε φορά που μιλάμε για τράπεζες μπερδεύομαι ιδεολογικά και θα σας εξηγήσω αμέσω γιατί. γιατί όταν άκουσα αυτά που είπε η κυρία Γκουλάρη μου θυμήσαν τον εαυτό μου. Εγώ είμαι συνήθω αυτός που υπερασπίζεται. Ε, ωστόσο, εδώ μιλάμε για υπεράσπιση τραπεζών και κάπως μπερδεύτηκα. Είμαι μισός Ιταλός, όπως ξέρετε, και δεν έχω αποφασίσει ακόμα για το ποια στάση θα τηρήσω. Όμως, εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συζητάμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ε, διασυνδεσιμότητα των ε, πολύ μεγάλων για να καταρρεύσουν πιστοτικών ιδρυμάτων. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και χωρίζονται στα δύο. Από τη μία υπάρχουν τροπολογίες που λένε ότι αν ε, κάνουμε υπερβολικές ρυθμίσεις θα σκοτώσουμε την οικονομία της αγοράς και δεν θα έχουμε αρκετή ρευστότητα στην αγορά. Και από την άλλη υπάρχει και μία δεύτερη αντιμετώπιση όπου θα μετατοπιστούν όλα τα προβλήματα στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα και μετά υπάρχουν συναντήσεις που λένε ότι δεν μπορείς να αγγίξεις αυτό το τραπεζικό σύστημα, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, γιατί θα πάνε όλα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει κίνδυνος μετά να χάσουμε στην Ευρώπη. Όμως, εγώ προσωπικά σε όλες τις ε, ακροάσεις που έχω παρευρεθεί για την ε, διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών δεν έχω ακούσει για το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην πραγματική οικονομία, δηλαδή τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Η χρηματοδότηση επενδύσεων δεν έχει να κάνει με το μέγεθος των τραπεζών ή την έλλειψη ρευστότητα. Πιστεύω πως το αντίθετο ισχύει μάλιστα, πως έχουμε ένα πρόβλημα με την ε, επέκταση των πιστώσεων με την ζήτηση και πιστεύω πως η ρύθμιση και η αντιμετώπιση των ε, τραπεζικών ιδρυμάτων που είναι πολύ μεγάλα για να καταρρεύσουν θα μας απελευθερώσουν κονδύλια για πραγματικές επενδύσεις. Τώρα, ως προς το που οδεύουμε, η Γκουε πιστεύει πως πρέπει να καθοριστούν σαφέστερα οι στόχοι στην αρχή μάλιστα της θητείας μας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα που είναι πάρα πολύ μεγάλα για να τα αφήσουμε να καταρρεύσουν. Υπάρχει το πρόβλημα των επιδοτήσεων, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά σε αυτό το χώρο. Πρέπει να αναφερθούν ρητά αυτή η στόχη στο σχέδιο έκθεση. Επίση πρέπει να ε, αναφερθούν όλες οι τράπεζες οι οποίες παρουσιάζουν συστημικούς κινδύνους με εξαίρεση όσους έχουν κάτω από 5% ασφάλεια ε, καταθέσεων. Εμείς ως Γκουε πάμε ακόμα παραπέρα και λέμε πως δεν χρειαζόμαστε μία μεγάλη δομή holding, διότι δεν θέλουμε να καταλήξουμε στα δικαστήρια με τους επόπτες μας, διότι σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες τράπεζες οι οποίες θα αμφισβητήσουν και θα υποβάλουν ένσταση σε αυτές τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Πολλές φορές και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. στο τέλο, ενδεχομένω να υπάρξει κάποιο συμβιβασμό με ένα σύστημα φωτεινού σηματοδότη ή κάτι παρόμοιο. Θα υπάρχουν λίγες κυρώσει για, ε, για την διαχείριση κεφαλαίων. Όμως αυτό που δεν θέλουμε να γίνει είναι να διακινδυνεύσει η εποπτεία και οι επόπτε. Τέλος. Θέλουμε να δοθεί ένα τέλος στην υπερβολική κερδοσκοπία και μια απαγόρευση των συναλλαγών με ίδια μέσα για να αποφευθούν οι αρνητικές συνέπειες στην πραγματική οικονομία. Και προσμένουμε την ανταλλαγή απόψεων και επίσης αναμένουμε να υπάρχει ένα αίσθημα υπευθυνότητας, διότι Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει με το χρέος, το κρατικό χρέος. Όλοι ξέρουμε τι έγινε με την Ελλάδα. Εκεί ο τραπεζικός τομέας δεν ήταν κατάλληλα, δεν είχε ε, κατάλληλο έλεγχο, κατάλληλα ρυθμισμένος. και δεν πρέπει να αφήσουμε τον τραπεζικό τομέα να γίνει ισχυρότερος από τα κράτη. Και η Google πραγματικά βρίσκεται στο πλευρό του φορολογούμενου. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ο Φίλιπ Λαμπέτς για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι το να παίρνει κανείς το λόγο μετά τον Γιάκοπ είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο βέβαια ε, αυτόν αλλά και άλλους. Ε, απλά σημείο προς σημείο στις παρατηρήσεις σας ε, εκφράστε αυτά που ήθελα να πω και εγώ και δεν θα τα επαναλάβω. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η ανθεκτικότητα μιας τράπεζας, καλύπτεται αυτό από το BRD, σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει τη συστημική ανθεκτικότητα. Ό,τι έχουμε κάνει με το BRD, δηλαδή διάβρωση βάση μεταφορά κερδών, But may not work in a με το BRD, συγγνώμη, το BEPS, ε, όλα αυτά αποσκοπούν στη συστημική ανθεκτικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι ελληνικέ τράπεζε είναι καταπληκτικέ και επενδυτικέ είναι κακέ και οι δύο, τα δύο δραστηριοτήτων είναι χρήσιμα. Έχουμε δει και ακούσει πολλά επιχειρήματα για το συνδυασμό των δύο των τραπεζών από την ίδια αυτή. Για να δημιουργήσουμε οικονομίε ε, εύρου και οικονομίε κλίμακα. Δεν το είδαμε όμω αυτό. Και από την άλλη πλευρά, το κόστο σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενο μετάδοση κινδύνων αρνητική μετάδοση. Νομίζω στο ΣΥΤΙ κάποιος το αυτό. Ότι πράγματι ε, πέρασε μια αρνητική νοοτροπία και στο retail banking. Αν λοιπόν δούμε μόνο τα αρνητικά και όχι τα θετικά από μια τέτοια συνύπαρξη, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να είναι αυτός ο στενός συνδυασμός των δύο επιλογή μας. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση. Εντάξει, ίσως τύπου φωτεινού σηματοδότη, δεν το λέμε έτσι Τροπολογίε τροπολογίες, αλλά τέλο μια προσέγγιση που να λέμε ότι πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο λέμε όχι στο συνδυασμό αυτών των δραστηριοτήτων υπό την ίδια στέγη. Αν οι δραστηριότητε τη Επενδυτική Τράπεζα είναι θεμητέ και νόμιμε, γιατί να μην ε, στέκονται αυτόνομα, με αυτονομία, χωρίς επιδότηση από τον κλάδο της λιανικής τραπεζικής, είτε άμεσα από το φορολογούμενο. Σε αυτήν την έννοια είμαι ακρεφνός φιλελεύθερος στην ε, πολιτική μου και στις απόψεις της αγορές. Αν δεν είναι οικονομικά βιώσιμη πολιτική και πρακτικέ μια επενδυτική τράπεζα, αυτό δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να επιβιώνει στην ε, οικονομία τη αγορά. Η τράπεζα που κάνει συναλλαγέ για ίδιο λογαριασμό πρέπει να διέπεται από διατάξει του Πογιάκου. Επίση, δεν διαφωνούμε τα εταιρικά, οι εταιρικοί θεσμοί ή οργανισμοί να πολλούν προϊόντα κάλυψης κινδύνων, όχι τα δικά τους όμως, προϊόντα που δημιουργούνται από άλλους. Άρα άλλοι φέρουν, ε, αναλαμβάνουν τον κίνδυνο και σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, νομίζω ότι όλες τις τράπεζες που χρησιμοποιούνται συστημικές θα πρέπει να τις περιλαμβάνουμε και γι' αυτό θα πρέπει να τρέξουμε στους εξετάμενου ορισμούς. Έχουμε ορισμό για το τι είναι βιώσιμο. Για ποια τράπεζα είναι βιώσιμη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού, Μηχανισμού. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον ορισμό διευρωπαϊκά και να χρησιμοποιήσουμε και τους ε, ορισμούς ε, του τέταρτου κανονισμού για την κεφαλαιακή επάρκεια. Γιατί τη διακριτική ευχαίρεια θέλω να πω δύο λέξει. Θα υπάρχει ένας βαθμός διακριτικής ευχαίρεια, περιορισμένο όμως. Πάλι ένα σύστημα φωτεινού σηματοδότη θα μπορούσε να λύσει τα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν. Αν πρέπει μπορεί εμπορική εντότητα κάπως να ξεχωριστεί. Όταν είναι κίτρινο το φως, ε, εκεί υπάρχει περιορισμένο περιθώριο λιγμών, αλλά πάντα στο όριο τη και πάνω από αυτά τα επίπεδα πράσινο, άρα δεν ισχύει ο κανονισμό, δεν καλύπτει τον σε αυτόν τον κανονισμό. Τεκτική ευχαίρεια προ του επόπτε. Μα δείχνει η εμπειρία μα ότι οι επόπτε έχουν τάση να έχουν μια σχέση συνενοχής κατά κάποιο τρόπο με τον επιβλέπον επιβλεπόμενο, τον εποπτευόμενο. Αυτό δεν είναι μια υγιή σχέση, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Αν δώσουμε λοιπόν μεγάλα περιθώρια δεκτικής ευχέρεια σε οργανισμούς που αποδεδειγμένα συνεργάζονται ε, αθέμητα με τους εποπτευόμενους, τότε τους δίνουμε προβολικά πολλές ε, αρμοδιότητες, άρα θα σε κίνδυνο με αυτόν τον τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον εντό Ευρωζώνη, τουλάχιστον Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι πιο απομακρυσμένη από πολιτική πλευρά τουλάχιστον από του εποπτευόμενου, άρα θα είναι πιο αυστηρή και αυτό θα κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Το βλέπουμε και με τι δράσει τη ΕΚΤ, ότι η ΕΚΤ συνεχώ προστατεύει το σύστημα των μεγάλων συστημικών τραπεζών. Ούτε μια φορά δεν έλαβε μια απόφαση που θα μπορούσε να θεωρηθεί αυστηρή από τις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Έχει πάρει όμως πολλές αποφάσεις που δεν θεωρήθηκαν αυστηρές από τα κρατημέλη για τα κατά κάποιο Να μην δώσουμε κυβερβολική δύναμη λοιπόν και στις κεντρικές τράπεζες. Uh, Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές ε, για ίδιο λογαριασμό, το prop trading πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τη χρηματοδότηση, παροχή πίστη εγγύσεων σε τέτοιους φορείς που κάνουν prop trading από την πίσω πόρτα. οι συναλλαγέ κρατικών ομολόγων ή ε, περιουσιακών στοιχείων ρευστότητα. Αυτό πρέπει να εξαιρεθεί. Να μην μπορούν δηλαδή να συναλλαστούν με τέτοια προϊόντα οι διάφοροι οργανισμοί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνετή διαχείριση κινδύνου τράπεζες που εκτίθενται και θα πρέπει να παρέχουν εξηγήσεις σε τακτά διαστήματα οι τράπεζες. Τι κάνουν με το prop trading και αν εκτίθενται σε κινδύνους. αν καλύπτεται, καλύπτονται οι συναλλαγές αυτές με κρατικά ομόλογα, κανένα πρόβλημα. Αν συναλλάσσονται όμως με κρατικά ομόλογα και δεν υπάρχει καμία σχέση προφανής με την έκθεσή του σε κίνδυνο, τότε αυτό είναι prop trading. Είναι συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό. Άρα θα πρέπει εκεί ο επόπτης να παρέμβει. Γιατί η συνθήκη προβλέπει συνετή διαχείριση κίνδυνων από Το οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Σε ό,τι το διαχωρισμό. Καλύτερα θα ήταν να έχουμε ένα είδος θετικού καταλόγου για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο prop trading και ότι δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο δεν είναι σημαντικό. Να μην ξεκινήσουμε με μαύρες λίστες, γκρίζες λίστες, αλλά με μια λευκή λίστα. Γιατί τις μαύρες λίστες πάντα κάτι ξεχνάμε. Για να δω τι άλλο θέλω να πω. Η Βρετανική εξαίρεση. Εγώ δεν είμαι Βρετανός υπήκος και έχω καταγραφεί να λέω ότι αν η διάταξη Vickers ε, καλύψει όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Ή και η ρύθμιση Λίκανεν επίση. Όχι, όχι, εμεί δεν θα το πετύχουμε. Αυτό το ξέρουμε, αλλά αυτό που προτείνουμε ω εναλλακτική λύση στην πρόταση τη Κομισιόν γιατί η διαχείριση εξαίρεση είναι όχι μια εξαίρεση για οποιαδήποτε χώρα, για κάθε χώρα, αλλά για τι τράπεζε οι οποίε ε, υπόκεινται σε ένα νομικό καθεστώ και φυσικά πρόκειται από μια χώρα, το οποίο καθεστώ σε ό,τι τον αντίκτυπο είναι ισοδύναμο με τα όσα προβλέπονται εδώ. Αυτό είναι μια λύση αν θέλουμε τις ε, νομικές ενστάσεις να τις υπερβούμε, τις εφτάσεις νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Θα περάσω στα γαλλικά για να απαντήσω στη Σιλβή. Συμφωνώ ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ακαιρότητα τη εσωτερική αγορά και συμφωνώ με τι ανησυχίε που εξέφρασε. Πράγματι, υπάρχει κίνδυνο. Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, να έχουμε πολλαπλασιασμό εθνικών ρυθμίσεων που όχι δεν θα περιορίσουν, αλλά θα αυξήσουν τον κατακαιρματισμό. Που είπε ότι ξεκίνησε με την κρίση του ευρώ και πολύ σωστά το μέρο των πρασίνων πρέπει να πω ότι με ενδιαφέρει καιρότητα τη αστέρικη αγορά. Η Βρετανική εξαίρεση δημιουργεί προβλήματα ω προ αυτό. Αν όμω καταφέρουμε με ευφυα να λύσουμε τα ζητήματα από κοινού, νομίζω θα το διαχειριστούμε το όλο αυτό θέμα. Εκεί που διαφοροποιούμε απέναντί σου, Σιλβί, και συμφωνώ με αυτά που είπε ο Φάμπιο, είναι ότι δεν έχουμε αποδείξει ότι μεγάλε συστημικέ τράπεζε που με τα περισσότερα του στοιχεία ε, συνεισφέρουν στην πραγματική οικονομία. Σε ένα βαθμό. Δεν βλέπω διαφορά με τις λέμικες τράπεζες. Οι τράπεζες που χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία αποκλειστικά και μέσω της κρίσης χρηματοδοτούν και στην διάρκεια της κρίσης μάλλον χρήμα συνέχισαν να χρηματοδοτούν και τους ΜΜΕ. αν έχει δημόσια εγγύηση μια τράπεζα γιατί συλλέγει φόρου, πράττει φόρου και μπορεί να ασχολείται μόνο με την πραγματική οικονομία, τότε όλα τα μέσα και όλο τον προπολογισμό θα τον αφιερώσει στην χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία, αλλά άρα δεν θα ασχοληθεί με δραστηριότητε αγορά. Που συχνά είναι πολύ αμφισβητήσιμο τι αποτέλεσμα έχουν για την πραγματική οικονομία. Και έχουμε ακούσει εκατομμύρια φορέ από το γαλλικό τραπεζικό τομέα η ίσως δραστηριότητα τη αγοράς σήμερα. Υπάρχει πολύ μεγάλος κατεκρεματισμός. Έχουμε πολλούς και μικρούς φορείς. Είχαμε την υπόθεση BMP, Παριμπά και σχετές Γενεράλ. Ακόμη και αν ίσχυε ο νόμος Glass-Steagall πάλι δεν θα είχαν λυθεί τα προβλήματα. και αν τις διαχωρίζαμε σε δύο κομμάτια θα εξαφανίζονταν. Και έχουμε και την Deutsche Bank που κατέχει μερίδια πολύ σημαντικά σε άλλες τράπεζες. Mm-hmm. Το θέμα είναι όλα αυτά τα σχόλια να οδηγήσουν σε επικοδομικές προτάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ Φιλίπ για την εκτενέστατη παρουσίασή σου. Μάρκο Τσάνι και την ομάδα EFTD. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς μια πρώτη θετική αποτίμηση διότι παρόλα αυτά η ποσότητα τροπολογιών, ο όγκος τροπολογιών για αυτό το τόσο σημαντική έκθεση είναι μια πρώτη θετική ένδειξη. Όλες οι ομάδες στο Κοινοβούλιο έχουν δώσει μεγάλη σημασία σε αυτήν την πρόταση. Είναι μια πρώτη θετική ένδειξη. Για να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Και όλοι μαζί να καταφέρουμε να βελτιώσουμε το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Δεν συμφωνώ καθόλου και δεν συμμερίζομαι καθόλου την αισιοδοξία του εισηγητού για τις συμβαστικές λύσεις. Βλέπω καταρχάς σε ορισμένα σημεία να υπάρχουν ε, αξεπέραστες δυσκολίες χάσμα μεταξύ των διαφορών πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Εύχομαι λοιπόν η αναζήτηση συμβαστικής επίλεσης, αυτός ο αγώνας με το ρολόι που δίνουμε, όπω είπαμε και συνάδελφοι προηγουμένως, γιατί το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί ω προς το θέμα αυτό. Δεν μπορεί παθητικά να περιμένει τη στάση του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, την έκφραση τους. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να μας καθυστερήσει να τοποθετηθούμε σε μια τελική έκφραση που δεν θα χρησιμεύσει σε τίποτα. Τώρα επί των τροπολογιών. Μετά από όσα άκουσα, Νομίζω όλοι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βασική προπόθεση. Εφόσον θέλουμε να διαθετήσουμε το χρηματοπιστωτικό τομέα, θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα ποιο είναι, για ποιου μιλάμε. Μιλάμε για πρόσωπα και οργανισμού και φορεί χωρί ενδιασμού ε, αδίστακτους που έχουν ε, παραποιήσει τα επιτόκια ε, τα, τις συναλλαγές, με το Lux LuxLeaks και την μεγάλη αυτή επενδυτική τράπεζα που χρηματοδοτούσε φοροφυγάδες, ατρομοκράτες επίσης. Να μην ξεχνάμε λοιπόν σε καμία περίπτωση με ποιους έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε αυστηρότατοι και να προτείνουμε κάτι, ένα νομοθέτημα που να είναι πολύ ισχυρό. Να μην αφήνει περιθώρια, να μην αφήνει δυνατότητες παρεμμηνίας και να έρχεται να βρει λύσεις στα κεντρικά σημεία που δημιουργούν πρόβλημα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για τη δική μου την ομάδα, τα σημαντικότατα αυτά ζητήματα που φαίνονται και στις τροπολογίες που προβάλαμε είναι τρία. Το too big to fail για τις τράπεζες. Και εδώ συμφωνώ ότι η διάσωση με ίδια μέσα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε περίπτωση συστημικής κρίσης. Πρέπει να αναλάβουμε δράση προτού προκύψει συστημική κρίση, δηλαδή πρέπει να την προλάβουμε. Η οδηγία για την εξηγήραση και τη διάσωση των τραπεζών αυτό που κάνει είναι να οριοθετήσει την κρίση μια συγκεκριμένη τράπεζα, όχι όμω μια συστημική κρίση. Αυτή δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Άρα πρέπει να αναζητήσουμε ένα σύνολο κανόνων που να είναι αποτελεσματικό κατά της διάστασης αυτής που όλο ένα και περισσότερο γίνεται συχνή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έπειτα, η διασύνδεση των τραπεζών μεταξύ τους, η παγκοσμιοποίηση σήμερα ουσιαστικά οδηγεί ένα μικρό λιθαράκι ενός μεγάλου ομίλου να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να δράσουμε ακριβώς ε, σε αυτό το σημείο. Να δούμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη διεθνή του διάσταση, το ευρωπαϊκό σύστημα να είναι πιο υγιές και να ε, είναι πιο κοντά στην πραγματική οικονομία και τις ανάγκες της. Και ένα τρίτο σημείο στο οποίο πρέπει να επιμείνω θέλω να ακουστεί και αυτό εδώ και θέλω να δώσουμε έμφαση είναι αυτό των παραγόγων. Διότι πράγματι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγόγων είναι τοξικά. Δεν έχουν καμία προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία. Είναι προϊόντα που προκύπτουν από κερδοσκοπικές ε, προθέσεις. Πρέπει λοιπόν και επ' αυτού να δράσουμε. Σε ό,τι αφορά το πεδίο του κανονισμού, και εγώ συμφωνώ απολύτω και υπέβαλα τροπολογίε από αυτή την έννοια. Ε, συμφωνώ να διευρυνθεί. Θα πρέπει να καλύψει τουλάχιστον όλε τι συστημικέ τράπεζε. Τι τράπεζε που, που, αφορά και ο ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Έπειτα, για το σύστημα αυτό κανόνων θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί και με τα, για τα κριτήρια ε, και να ακολουθήσουμε ίσω τον απλούστερο δρόμο, αλλά που είναι και αποτελεσματικότερος, της ε, σαφούς απλής νομοθεσίας. Ορίζουμε κριτήρια, παραμέτρους για τον κίνδυνο με δύο-τρία σημεία που θα λένε ποιοι είναι οι παράγοντε κινδύνου, οι μεγαλύτεροι παράγοντες κινδύνου για τους συλλογισμού των τραπεζών. Και αν βασιστούμε σε αυτά τα κριτήρια, θα μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα διαχωρισμό υποχρεωτικό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να αφήσουμε στην διακριτική ευχέρεια, στην υπέρμετρη διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρχών, το διαχωρισμό. Θα συμφωνήσω εδώ απολύτω με αυτό που έλεγε ο Φίλιπ Λάμπερτ. Σε μερικέ περιπτώσει υπάρχουν συγκρούσει συμφερόντων, ε, υπάρχουν καταστάσει ιδιαίτερα σαφεί ε, και πολύ αδιαφανεί. και στην Ιταλία το είδαμε και αυτό, και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Θα πρέπει λοιπόν να ε, κοιτάξουμε να μην επιτραπεί τέτοια χαλαρότητα. Και κατά τα άλλα, ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε κάποια συμβαστική λύση, αλλά τέτοια συμβαστική λύση που να βελτιώνει πραγματικά το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε. Μια μικρή διαδικασία, κάτι Μετά η Κομισιόν και μετά η Συγητή σε έναν εγώ στον κατάλογο των μιλών, ο κύριο Βάλτ. Και αν με πρέπει να κλείσω τώρα τον κατάλογο, αν δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει το λόγο που δεν βλέπω, ο συνάδελφο Βάλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σίμων. Θα είμαι λίγο σύντομο για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συγκεκριτής μας να κάνουν μια σύνοψη. Πήραμε τις τροπολογίες και νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε. Και πραγματικά ο κύριος Χόκμαρκ μας ε, έδωσε μια εξαιρετική βάση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ε, για το πώς θα συνεχίσουμε. Πιστεύω πως οι τροπολογίες έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι απέχουμε πάρα πολύ από το να συμφωνήσουμε. Ωστόσο, συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή και στηρίζω απόλυτα την ε, εκτίμησή του για το, την επίλυση μέσω των κινδύνων. Χρειάζεται να μειωθεί ο κίνδυνος που προκύπτει από ορισμένε εμπορικές δραστηριότητες και δεν ε, θα γίνει αυτό απαραίτητα με αυτόν τον διαχωρισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, να πω ότι αμφιβάλλω για το αν ένας αυτόματος διαχωρισμός θα επηρεάσει ή θα αλλάξει τα πράγματα. Πιστεύω πως, μια, πως ένας αυτόματος διαχωρισμός θα πρέπει να παραμένει ένα μέτρο τελευταίας λύσης. Επίσης, είμαι πεπισμένος ότι στο μέλλον πρέπει να στοχεύσουμε σε, μια, σε ένα θεματολόγιο ανάπτυξης για την Ευρώπη. Πιστεύω, ε, ξέρω πως υπάρχουν αρκετοί από εσάς οι οποίοι υποστηρίζουν και την ανάπτυξη και ε, προώθηση των επενδύσεων και ταυτόχρονα έναν διαχωρισμό από τις ε, καθολικές τράπεζες. Πιστεύω πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να έχουν ξανά τη δυνατότητα να παρέχουν ρευστότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ σωστό. Όμως, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα οι τράπεζες θα πρέπει ταυτόχρονα να παρέχουν ρευστότητα, πιστοτική ρευστότητα για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διάθεσης τίτλων στην αγορά ε, περιουσιακών στοιχείων. Στην αγορά αξιών, με συγχωρείτε. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε με το εναλλακτικό ταμείο επενδύσεων. Πιστεύω πως ε, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία χρειάζονται στρατηγικές επενδύσεις. Υπάρχει ρύθμιση μέσω οδηγίας αυτού του Ταμείου Επενδύσεων και αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι να διασφαλιστεί η ε, συνεκτικότητα μεταξύ των οδηγιών. Επίσης, προσανατολίστηκα στο γερμανικό σύστημα διαχωρισμού των τραπεζών στις δικές μου τροπολογίες, οι οποίες δεν προβλέπουν αυτού του είδους τη μόχλεση και επίσης ε, αποκλείονται οι επενδυτικές τράπεζες από κάθε είδους εμπορικές ε, συναλλαγές. Επίσης, πιστεύω πως με τις τροπολογίες που έχω υποβάλει φαίνεται ξεκάθαρα το πόση δουλειά έχουμε μπροστά μας. Όπως, όπως είπα, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στον εισηγητή όσο και στους κοιόδης εισηγητές για το ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να έχουμε μια σωστή και συνετή λύση. Δεν θα είναι εύκολο, είναι όμως εφικτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλτ. Δεν θέλω να αφήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Προϋπολογισμού να περιμένουν πάρα πολύ έξω από την αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον κύριο Μάρτιν Σπότ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή καλωσορίζει την πρόταση του εισηγητού του κύριου Χέκμαρκ, καθώς και τις πολυάριθμες τροπολογίες. Και η έκθεση και οι τροπολογίες είναι μια πολύ καλή βάση για την συνέχιση των συζητήσεών μας και για να επιτελέσουμε πρόοδο. Προβλέπουν μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία για την όλη μελέτη του θέματος. Δε, συμφωνούμε με την έμφαση που δίνει ο συζητητής και πολλοί συναδελφοί του για την ανάγκη εξέβρεση σωστή σημείου ισορροπίας μεταξύ αντιμετώπισης των κινδύνων που παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλες τράπεζες, μεγάλη τραπεζική όμιλη too big to fail, αλλά και το να μην εμποδίσουμε τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας από την άλλη. Παρόλο που υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ ανάγκε από τι δύο πλευρέ, η Επιτροπή, όπω και η Ευρωβουλευτή κυρία Γκουλάρ, θεωρεί ότι είναι εφικτό να βρούμε ένα ε, έδαφο συνεννόηση και να καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει. Γι' αυτό είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι προσπάθειε καταβάλει και η Λατωνική Προεδρία στο Συμβούλιο με συγκεκριμένη πρόταση επιτάπητος ε, που είναι πολλά υποσχόμενη. Παραμένουμε στη διάθεση του συγητού και όλων των υπολείπων ε, μελών αυτής της Επιτροπής για να βρούμε μια πραγματική και εφικτή λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εισηγητής μας κύριος Χότμαρ έχει τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για, αυτές τις, ε, για αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Καλωσορίζουμε Καλωσορίζω τι προτάσει όλων, γιατί μην ξεχνάμε ότι μόλι μιλάμε για διαθέτηση των τραπεζών, όλοι αρχίζουν να ακούγονται φιλελεύθεροι ω προ τι τράπεζε. Όλοι έρχονται και λένε είμαι φιλελεύθερο για την αγορά των τραπεζών. Το καλωσορίζω, αυτό είναι ευχάριστο. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο σαφής βέβαια και ο Γιάκομπ ως προς αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ε, να πω το εξή. Και αυτό έχει συνέπειες για όλα όσα κάνουμε. Για μας που ούτως ή άλλως παραδοσιακά πιστεύαμε στην οικονομία της αγοράς, ένα πράγμα είναι σαφές. Η οικονομία της αγοράς δεν είναι πανάκια. Πρέπει να υπάρχει ισχυρό κράτος είναι ενδιαφέρον όταν το συζητήσαμε και κιόλα με την αφορμή τη οδηγία για την εξηγία των τραπεζών. Ήμουν και τότε σαφή όταν το συζητούσαμε. Ε, η διάδοση με τα ίδια μέσα δεν είναι λύση για όλα. Και το λέω και το δηλώνω. Κάποιε φορέ αισθάνθηκα πολύ μεγάλη μοναξιά όταν το υποστήριζα αυτό. Διότι σχεδόν όλοι σε αυτή την επιτροπή από την αρχή έλεγαν ότι το bail-in, η διάδοση με ίδια μέσα, είναι η λύση. Και Επαναλάμβανοντα σχεδόν αυτά που είπαν ο Φάμπιο και ο Φιλίπ μόλι τώρα. Στι συστημικές κρίσεις, και ήταν ε, και η Λίσα, η Ελίζα τότε παρούσα, δεν αφορά μόνο την σωστή ισορροπία στην οικονομία. Γι' αυτό η οδηγία για την αξία των τραπεζών μας έδειξε ένα δρόμο επιθέβεσης λύσης. Τα επικίνδυνα χρέη είναι το θέμα. Ε, το, ο 80% του bail-in στην περίπτωση συστημική κρίσης μπορεί να αποτιμηθεί σωστά. Αλλά πρέπει να μην παραβλέπουμε την οδηγία για την εξυγίανση λέγοντα εντάξει αυτό τώρα έγινε, πέρασε και το ξεχνάμε. Όχι. Ε, για την ασφαλεία των επενδυτών η Επιτροπή μα έχει επενδύσει πολλά για να υπάρξει σωστή εποπτεία στην Ευρώπη σε διαφορετικά επίπεδα. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα το κάναμε αυτό αθώα γιατί δεν του έχουμε εμπιστοσύνη. Θα πρέπει, πολύ να, θα πρέπει να ξαναδουλέψουμε πολλά πράγματα αν το αποθετηθούμε έτσι. Αυτό που θέλουμε είναι οι επόπτες να έχουν το καλύτερο σύστημα εργαλείων. Όχι μόνο για το τι θα κάνουν, αλλά η διαφάνεια να λειτουργεί και για αυτούς ως εργαλείο, για να μπορούν να δουν τα προβλήματα, να τα εξετάσουν, αλλά και για να υπάρχει διαφάνεια και για το κοινό. Θα ήθελα και θα πάψω εδώ, γιατί ξέρω ότι έχουμε και συζήτηση για το στρατηγικό ταμείο. Θα ήθελα να είμαστε λίγο θετικότεροι. Διότι άμα ακούσω κάτι συναδέλφους που λένε ότι δεν είμαστε αισιόδοξοι για τις συμβαστικές λύσεις, γιατί ο καθένας έχει τις απόψεις του και εγώ τις δικές μου, δίκιο έχουν, ε, τι να σας πω, πάντοτε θεωρώ τις απόψεις μου σωστές, αλλιώς θα τις είχα. αλλά, αλλά έδειξε έναν δρόμο για την εξέβρεση λύσεων. Και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, και εμείς και άλλες, Γιώργ, πρέπει να βρούμε τη λύση για να έχουμε μια νομοθεσία, ένα νομοθέτημα. Επιτρέπουμε στον άλλον να έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι και αυτός έχει δίκιο. Γι' αυτό ε, είπα ότι θα πρέπει να υπερβούμε τις, τα σημεία διαφωνίας, ε, ακολουθώντας μια νέα προσέγγιση για τον παράγοντα της διαφάνειας. Ίσως ε, ήταν πολύ ιστορική η σκοπιά μου όταν μίλησα για, τη, για τα βενετσιάνικα παράθυρα ή τις βενετσιάνικες θύρες, αλλά οι σοσιαλιστές ε, ε, άκουσα από πριν από τον Γιάκοπο ότι είσαστε πρόθυμοι να συμβαστείτε. Νομίζω οι συζητήσεις μας έχουν πάρει τη σωστή κατεύθυνση. Εν τέλει, Πρόεδρε, Είμαι αισιόδοξο. Είμαι αισιόδοξο και βλέπετε ότι είναι 17 και 30 αυτή τη στιγμή. Άρα είναι ακριβώ η ώρα μου να σταματήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γκούναρ, και ευχαριστώ πολύ που πραγματικά κράτησε τα χρονικά όρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου εσά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα. Να σα πω πολύ σύντομα ότι η ψηφοφορία προβλέπεται για τι 23 Μαρτίου και ο ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Επίση να σα ε, ε, υπενθυμίσω ότι υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δύο ψηφοφορίες και να σας ευχαριστήσω στο τέλο για ε, την συνεδρίαση. Θα αρχίσει τώρα η κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Oh.